Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες μου και κύριοι, ας αρχίσουμε. For this afternoon. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε. Thank you for coming. Not many of us. Πρώτον, ευχαριστίες που ήρθατε. Είναι μικρή με, ναι, η εκπροσώπηση, αλλά πάρα πολύ σημαντική και παρακαλώ να παραμείνετε και να μην φύγετε πριν τις 6.30. Ε, αν μου επιτρέπετε να σας το ζητήσω. Λοιπόν, Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου 2015, 3 με 6.30. Is included in the... Ε, έχετε την ημερήσια διάταξή σας, το σχέδιο συγκεκριμένα και θα σας πρότεινα μερικές αλλαγές. τα σημεία 7 και 14 αλλάζουν μεταξύ τους. Ο εισηγητής Λεβαντόφσκι για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα συζητηθεί το θέμα του 9 με 10 αύριο το πρωί και οι συντονιστές θα είναι το τελευταίο αυριανό θέμα από τις 5 μέχρι τα 6.30. Δηλαδή αλλάζει η συνεδρίαση των συντονιστών με τον κύριο Λεβαντόφσκι. Καλά, δεν είναι και καμιά τραγική αλλαγή αυτή. Λοιπόν, σημείο 8 ή στα 2 ψηφοφορία σύμφωνα με τον κανόνα, το άρθρο 73.5 του κανονισμού του συναδέλφου Τζορίνιο αναβλήθηκε αυτό το θέμα για τις 13 Οκτωβρίου 2015 γιατί συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Και το ε, σημείο 7α προστίθεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά αυτά που σας είπα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι τρεις αλλαγές. Οι συντονιστές ασχολούνται με την αναθεώρηση του τρόπου που ανατίθενται εκθέσεις και οι γνωμοδοτήσεις κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών την περασμένη εβδομάδα ελήφθη αυτή η θέση. Με μια επιστολή της 17ης ε, ενάτου οι συντονιστές των ΓΚΟΕ, Πρασίνων και η FTT ζήτησαν να τεθεί σε ψηφοφορία η θέση αυτή στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας. Βάσει της επιστολής αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 205 του κανονισμού που έχει τη σημασία του αυτό. Υπάρχει και τέτοιος κανονισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει σχετικό άρθρο λοιπόν. Θα ψηφίσουμε την απόφαση των συντονιστών για την ανάθεση των εκθέσεων όπως ζητούν με την επιστολή τους οι συντονιστές που σας ανέφερα. Συμφωνείτε? Δηλαδή για να δούμε αν την υπερψηφίζει η Ολομέλεια της Επιτροπής ή την καταψηφίζουμε. Την απόφαση αυτή των συντονιστών. Στις 10 η ώρα αύριο θα γίνει αυτό. Πρόκειται για την απόφαση σχετικά με τον τρόπο που ανατίθεται και διανέμονται οι εκθέσεις και οι γνωμοδοτήσεις. Στις 15 του συνεδρίασαν οι συντονιστές. Αυτά είναι βάση του άρθρου 205 του κανονισμού και το ζήτησαν με επιστολή τους η ΓΚΟΕ, η Πράσινη και η FTD. Τρεις πολιτικές ομάδες. Βεβαίω το κείμενο θα διανυμηθεί σε όλα τα μέλη αυτή τη στιγμή εγκριθεί. Ο κατάλογος ψηφοφορίας. Λοιπόν, τρεις προτάσεις έχουμε. Έχετε ερωτήσει σχετικά με την ημέρησια διάταξη. Ο κύριος Ρόιλ, παρακαλώ. Μια στιγμή να βάλω και κανένα ακουστικό. Well, well. I ready. Okay, then I can start. Yeah. Ναι. Λοιπόν, έχω μια συμπληρωματική ερώτηση, διευκρινιστική, για το πώς αναστήθενται οι εκθέσεις. Αυτό ήταν στο παρελθόν πάντα κάτι το οποίο το αποφάσισαν και το κανόνιζαν οι συντονιστέ. Αυτό είναι ειδική δουλειά και καθήκον των συντονιστών. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί αλλάζει και είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί αν στο μέλλον ε, αρχίζουμε να ψηφίζουμε όλα τα διαδικαστικά, τότε θα το κάνω και για δικά μου θέματα που με ενδιαφέρουν εμένα. Λοιπόν, είτε αυτό είναι δουλειά των συντονιστών και την κάνουν, να την κάνουν πάντα, είτε θα τα αλλάξουμε και στο μέλλον θα ισχύει αυτό και για άλλα θέματα. Αν κάποια πολιτική ομάδα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέλημα, να το φέρνει στην Ολομέλεια της Επιτροπής να το ψηφίζει. Αν ε, ε, εγκρίνουμε αλλαγές στο σύστημα ανάθεσης των εκθέσεων, αυτό στο μέλλον θα γίνεται πάντα με τους συντονιστές, όχι από την Επιτροπή. Αυτό που ψηφίζουμε είναι αν θα αλλάξει το σύστημα με το οποίο μοιράζουμε τις εκθέσεις. Όχι τον κανόνα ότι ε, ευθύνονται για την κατανομή οι ε, συντονιστές. Αυτό δεν αλλάζει. Παραμένει αρμοδιότητα και καθήκον των συντονιστών. Αυτό που θα ψηφίσουμε είναι αν θα αλλάξουμε το σύστημα, τον τρόπο. Το σύστημα με το οποίο μοιράζονται οι εκθέσεις και το έχουν ζητήσει τρεις πολιτικές ομάδες να το αποφασίσει αυτό η Επιτροπή μας και όχι οι συντονιστέ. Εντάξει. Παραμένει όμως η απόφαση ουσιαστική στα χέρια των συντονιστών για το πώ θα μοιράζονται οι εκθέσεις. Συνάδελφοι, είναι σαφέ νομίζω αυτό. Δεν ξέρω. Κύριε Ρόελ, ε, το καταλάβατε. Ναι, το είχα καταλάβει και από πριν, μην ανησυχείτε. Ε, το τι ψηφίζουμε, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ο κανόνας που ίσχυε μέχρι τώρα ε, πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν έχει αποφασίσει η Επιτροπή. Οι συντονιστές την είχαν αποφασίσει πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι. Και εάν αυτό πια δεν το αποφασίζουν οι συντονιστές αλλά το σύνολο της Επιτροπής, ήθελα να σας πω ότι και στο μέλλον οτιδήποτε έχει να κάνει με κανόνες θα πρέπει να έρχονται να ψηφίζονται στην Επιτροπή. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό άπαξ. Όχι, αγαπητέ συνάδελφε, Άλμπερτ, λέει ο πρόεδρος. Δεν υπήρχε έτοιμα να ψηφιστεί αυτό στην Επιτροπή προηγουμένως. Ποτέ δεν το έχει ζητήσει κανένας. Όλες οι αποφάσεις των συντονιστών ίσχυαν. Αυτή τη φορά ζητήθηκε από τρεις πολιτικές ομάδες να το τσεκάρουμε στην Επιτροπή. Είναι έκτακτη η περίσταση και ασυνήθιστη μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εάν όμως το ζητήσουν τρεις πολιτικές ομάδες που δικαιούνται, η υποχρέωση είμαι να συζητήσω να ψηφίσετε για τίποτα άλλο. Είναι τελείως έκτακτη και συνήθιστη η περίσταση. Στο παρελθόν κανείς. Όταν εσύ προέδρευες ας πούμε στην Επιτροπή, κανείς δεν το είχε ζητήσει αυτό ποτέ, να γίνει έλεγχος στην Επιτροπή. Αλλά στην αρχή των συνεδριάσεων, κάθε φορά μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών, ανακοινώνω τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Έτσι δεν είναι για πολλά θέματα. Και αν έχετε καμιά αντίρρηση, το λέτε και σας ζητάω να εκφράζεστε. Και συνήθως κανείς δεν έχει αντίρρηση. Δεν αλλάζουμε τίποτα λοιπόν σε σχέση με όλα αυτά. Ε, τώρα αν πρέπει οπωσδήποτε να το αρχίσει η συζήτηση μπορώ να το κάνω. Ε, ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, όχι. Ο κύριος Ηλικιώτη, θέλετε να πείτε τίποτα. Ε, ναι, Πρόεδρε, απλώ πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι η διαδικασία και αποφασίζουν τι εκθέσει και το διαμερισμό στου συντονιστέ. Όμω, γιατί νιώσαμε την ανάγκη να θέσουμε το θέμα στην Επιτροπή. Γιατί αλλάζει το σύστημα, ε, όχι στην αρχή όπω αποφασίζεται πάντα, κατά τη διάρκεια που είμαστε σε αυτήν την περίοδο. Δηλαδή, αν αυτή η πρόταση ερχόταν για παράδειγμα όταν θα υπάρχει το midterm και υπάρχει μια συζήτηση εμείς θεωρούμε επειδή αυτό αλλάζει ξαφνικά θεωρούσαμε ότι πιο σωστό ότι να γίνει συζήτηση και ψηφορία εδώ στην Επιτροπή μια και υπάρχει αυτή η μεγάλη διάσταση στι απόψει μεταξύ των συντονιστών ε, χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία του θέματος. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συντονιστές, Υποθέτω ότι μπορείτε να ενημερώσετε τα μέλη των ομάδων σας για την κατάσταση όπως έχει. Γιατί κανονικά θα πρέπει να αποφεύγονται συζητήσεις. Έχουμε ψηφοφορίες αύριο, όχι μακρά συζήτηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Η ψηφοφορία είναι ψηφοφορία. Αύριο το πρωί έχουμε ψηφοφορίες. Λοιπόν, θα παρακαλούσα όλους τους συντονιστές να ενημερώσουν τα μέλη των πολιτικών τους ομάδων σχετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αν θέλουμε αύριο να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και προχωρούμε. Σας ερωτώ λοιπόν, αυτές τις αλλαγές δέχεστε την ημερήσια διάταξη μπορεί να εγκριθεί με τις τρεις αυτές αλλαγές που πρότεινα. Ωραία, δεν διαφωνεί κανείς. Ανακοινώσει του Προέδρου. Συνεδρίασε το μάλλον θα συνεδριάσει διευρυγμένο Προεδρείο στο Στρασβούργο για την Ενεργειακή Ένωση στις 6 Οκτωβρίου του 2015 παρουσία του Αντιπροέδρου Σεύσκοβιτς 8.30 με 10 το βράδυ στην αίθουσα Winston Churchill Week 200. Άτυπη συζήτηση με τον κύριο Σεύσκοβιτς στο Διευρυμένο Προεδρείο. 6 Οκτωβρίου, 8.30 με 10 το βράδυ. Θα έχουμε τον Αντιπρόεδρο Σεύσκοβιτς και τα μέλη της Επιτροπής μας πάρα πολύ σημαντική συζήτηση άτυπη. Το έχουμε ξανακάνει αυτό με άλλο επίτροπο. ήταν. ήτανε. Α, ο επίτροπο Μοέντα. Πρόσφατα. Ε, ε. Με τον ε, επίτροπο Μοέντα. τρία, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που βλέπετε, 15-16 Ιουλίου 2015. Έχετε τα πρακτικά στα χέρια σας. Εάν δεν έχετε άλλα σχόλια θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο. Ωραία. Σημείο 4. Ορίζον 2020. Πρώτα αποτελέσματα ανταλλαγή απόψεων με τον Ρόμπερτ Γιάν Σμιτ, Γενικό Διευθυντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε πολύ συχνά προσκεκλημένος μας κύριε Γενική Διευθυντά. Είστε προσφυλής και οικείος ε, της Επιτροπής. Καλώς ορίσατε. Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν, πρώτα αποτελέσματα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ορίζον 2020. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Γενική Διευθυντά ότι και ο Επίτροπος Μοέντας είναι σε μόνιμη επαφή με την ε, Επιτροπή μας και τα μέλη της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε διερώς ενήμεροι για τα τεκτενόμενα Διότι όπως γνωρίζουμε η πολιτική καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα κτλ. είναι καθημερινό μας μέλημα. Να μην σας πω και τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2000, από τα σημαντικότερα. Ε, και ε, μη τι άλλο και επιτέλους πρέπει να πετύχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό μετά από 15 χρόνια. Πολιτικής καινοτομίας. Στην Ευρώπη 2020 παντού. Στρατηγική της Λισαβόνας όλα αυτά έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε κάποια στιγμή θα πρέπει να πετύχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα τα καταφέρουμε. Ιδού το ερώτημα. Και είστε και διευθυντής εσείς γενικός εδώ και πολλά χρόνια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου προσφέρετε την ε, δυνατότητα να είμαι σήμερα μαζί σας, ώστε να σας ενημερώσω για τα πρώτα αποτελέσματα του Horizon 2020. Μάλιστα, ο Επίτροπος μου έδωσε, σας έστειλε ήδη λεπτομερείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που υποβάλλατε, ωστόσο, ε, οπότε μάλλον δεν θα μπω σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να εστιάσω την σύντομη μου εισήγηση Καταρχάς, στο πού βρισκόμαστε με τον ορίζοντα 2020 και πόσο αποδίδουμε στις βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Γιατί θυμάστε ότι όταν είχαμε στις διαπραγματεύσεις είχατε κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και θα σας πω, θα σας ενημερώσω τι κάνουμε για αυτά τα θέματα τα οποία θεωρείται πολύ σημαντικά. Θα σας μιλήσω για τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα, αλλά δεν θα διστάσω να σας ε, αναφέρω κάποιες ανησυχίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν να αρχίσω με τις επιτυχίες. Ο ορίζοντας 2020 είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει 65.000 προτάσεις. Αυτό δείχνει ότι πάρα πολλοί ετούντες βρίσκουν το δρόμο τους προς τα προγράμματα των Βρυξελών. Εν γέννη, η ποιότητα αυτών των προτάσεων που λαμβάνουμε είναι καλή. Σας έχουμε στείλει, θα δείτε μπροστά σας αυτό το, το βιβλιαράκι που δεν περιλαμβάνει ακόμα όλες τις 65.000 προτάσεις γιατί αρκετές από αυτές ακόμα είναι στην αξιολόγηση αλλά αντικατοπτρίζει ποια είναι η μοίρα των 31.000 προτάσεων που έχουμε ήδη εξετάσει. Βλέπουμε σαφώς ότι οι ετούντες ε, βρίσκουν θετική τη νέα προσέγγιση ε, που εστιάζει στις βασικές κοινωνιακές ε, προκλήσεις, βλέπουν, βλέπουν το μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής και τα προσιτά και κατανοητά κριτήρια. Αυτά ήταν τα σημεία που θέλατε να δείτε εσείς. Και κάτι ακόμα που κατά δεύτερο λόγο τονίσατε πολύ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εδώ, ε, σε αυτή την Επιτροπή, είπατε ότι δεν θέλετε να έχουμε ένα κλειστό ε, πρόγραμμα. 40% των ετούντων είναι καινούργοι, πρέπει να σας πω. Ε, και από αυτούς του 40% το 80% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ακριβώς αυτό μας είχατε ζητήσει, να μην έχουμε κλειστά ε, ε, κλειστό κύκλωμα ε, και να έχουμε νέες επιχειρήσεις. Τώρα, κάτι ακόμα που σχετίζεται και είναι επιτυχία και σχετίζεται με την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χάρη στο μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νεότευτων επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων. Ε, το 25% του προπολογισμού των πυλώνων 2 και 3 ε, θα πρέπει να αφιερωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως σήμερα βρισκόμαστε στο 23%. Δηλαδή θα ξεπεράσουμε τους στόχους και αυτό είναι πολύ καλό νέο για την κυρία Τόγια και τον Παόλο Ρούπιχ που ιδιαίτερα επέμειναν για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέταρτη μου παρατήρηση ε, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ε, παρακαθήμενό μου πρόεδρο, αλλά και ο κύριος Τούρμες ζητούσε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες ε, για την ενέργεια. Η ενέργεια στη διάρκεια των διπροματεύσεων ήταν το κεντρικό ζήτημα το κεντρικό ε, θέμα που μας απασχόλησε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση που θα δινόταν στην έρευνα για τα μη στερεά και την ε, ενημέρωση για τον εξυγχρονισμό της αγοράς. Το 85% του προϋπολογισμού λοιπόν έπρεπε να δαπανηθεί στις ανανεώσιμες και το 15% στην ε, νέα αγορά. Για τα μη στερεά είμαστε τώρα στο 90%. Ε, πετυχαίνουμε λοιπόν τους ε, ε, στόχους μας κατά το 90% αυτή τη στιγμή. Σημείο 5. Η Αρσή. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που κάναμε ποτέ για την Ευρωπαϊκή Επιστήμη είναι η δημιουργία του ERC. Είχαμε, είδα, είχαμε διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος γνωρίζει πόσο επιτυχές είναι αυτό το κέντρο, διότι έχει αποτελέσει πλέον ε, παγκόσμια προδιαγραφή η έκθεσή του και προκαλεί ε, ε, ενδιαφέρον από ολόκληρο τον κόσμο. Να σας πω ότι βέβαια ένας άνθρωπος ήταν πολύ σημαντικός και ήταν η Αντζέλικα Νίμπλερ που τότε έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στην θέσπιση αυτού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου. Ε, θέλω να την ευχαριστήσω λοιπόν ε, ιδιαίτερος, αλλά και σας Πρόεδρε που από την πρώτη μέρα υποστηρίξατε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού ε, Ερευνητικού Συμβουλίου. Κρίσιν Έλερ, που μόλις βγήκε. Fast track για την καινοτομία. γιατί Ήταν το πρώτο σημείο που και το πιο σημαντικό που ήθελε να μπει στον, ορα, ορίζοντα 2020 και είμαι ευτυχή που αυτή η νέα πρωτοβουλία για την οποία στην αρχή ήμασταν κάπως διστακτικοί είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έχουμε δηλαδή 264 προτάσεις ενώ μπορούμε να επιλέξουμε μόνο 16. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο τεράστιο είναι το ενδιαφέρον για αυτή την πιλωτική δράση γιατί ακόμα είναι πιλωτική η δράση αυτή και σίγουρα θα είναι ε, ε, σε όλες οι προτάσεις και η ποιότητά τους. Ε, σημείο 7. Η διάδοση της αριστείας και η διεύρυνση της συμμετοχής. Βλέπω τον κύριο Ρόιλ που κάθεται εδώ που μαζί με την κυρία Κουντρίτσκα ζήτησαν τη διεύρυνση των πρωτοβουλειών, τη δημιουργία ομάδων, την μοιρασία του κόστους και εδώ και ο Πρόεδρος επέμεινε και έχουμε δει τεράστιο ενδιαφέρον ε, όσον αφορά τις αιτήσει. Για μένα όμως η πιο μεγάλη επιτυχία του Horizon 2020 και είναι το τελευταίο μου σημείο είναι το 8, είναι η απλοποίηση. Η απλοποίηση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά με το παρελθόν. Και είμαι ευγνώμων προς την Επιτροπή σας γιατί εδώ παίξατε πολύ κρίσιμο ρόλο ε, κύριος Καρβάλιο με ιδιαίτερη έκθεσή του με 54 απλουστευτικά μέτρα ε, μας ε, επέτρεψε να απλοποιήσουμε το πρόγραμμα και είμαστε γνώμονες για την επιμονή αυτή και έτσι μπορέσαμε όχι μόνο να μιλήσουμε αλλά και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές. Τώρα, ανησυχίες έχω επίσης που επίσης θα τις μοιραστώ μαζί σας κατέστησα σαφές ότι ε, όσον αφορά τις προτεραιότητές σας έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και ότι είναι πολύ δημοφιλές το Horizon 2020. Αλλά υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Καταρχήν, πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της Ένωσης. Έχουμε στην Ευρώπη ένα χάσμα καινοτομίας και επιστήμης, αλλά πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην διευρυνθεί περισσότερο. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του ορίζοντα 2020 δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, αλλά χρειάζεται να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Και βεβαίως υπάρχουν ε, συνέργειες ανάμεσα στο ορίζον 2020 και τα διευθυντικά ταμεία και είναι πολύ ουσιαστικές. Και είχαμε μια συνάντηση με. Μάλλον σύντομα θα έχω μια συνάντηση με τον κύριο Βανίστερ εδώ για να το συζητήσουμε αυτό με κάθε λεπτομέρεια. Δεύτερο σημείο είναι η διεθνή συμμετοχή. Ο Horizon 2020 είναι ανοιχτό για ολόκληρο τον κόσμο. Και θα πρέπει πολύ περισσότερο από ποτέ να συνδεθούμε με του ε, έξυπνους ε, Αμερικανούς, Κινέζους, Βραζιλιάνους προς το δικό μας συμφέρον. Εμείς παράγουμε το 1 τρίτο της γνώσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά είναι σαφές ότι η παγκόσμια γνώση διαρκώς όλο ένα και περισσότερο ε, δημιουργείται εκτός Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να συνδεόμαστε με τα καλύτερα μυαλά όπου και αν βρίσκονται και θα ήθελα να δω πολύ περισσότερη διεθνή ε, συμμετοχή στο Horizon 2020. Κάτι ακόμα που μας απασχολεί είναι η απλοποίηση η δουλειά αυτή ποτέ δεν τελειώνει, όπως έχει πει και ο Επίτροπος Μοέδας. Ήδη αυτή την εβδομάδα διοργανώνουμε ένα τεράστιο σεμινάριο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετέχουν για να δουν πώς ακόμα περισσότερο μπορούμε να απλοποιήσουμε. Έχουμε, θα ξεκινήσουμε online διαβούλευση και θα είναι κάτι που θα βρίσκεται συνέχεια στην ημερησία μας διάταξη. Αν όμως, Πρόεδρε, με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία αυτή τη στιγμή, θα είμαι ειλικρινής είναι η υπερβολική ε, συμμετοχή. Έχουμε πλημμυρίσει από τις προτάσεις ε, και το ποσοστό επιτυχίας είναι 12 με 14% ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν, 14, ε, ήταν 20%. Πρέπει να απορρίψουμε πολλές προτάσεις. Έχει, υπάρχει τεράστια δημιουργικότητα και δυνατότητα καινοτομία στην μας. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται να απορρίπτουμε σε τεράστιο ποσοστό. Και αυτό που δεικνύει, Πρόεδρε, ένα πράγμα που είναι δύσκολο να το δεχτούμε, ότι εσείς και η Επιτροπή σας και αυτό το Κοινοβούλιο είχατε δίκιο όταν είπατε ότι ο προπολογισμό του Horizon 2020 ε, θα πρέπει να είναι 100 δις και όχι, και όχι 80. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Καρβάλιο, πρώην Ευρωβουλευτής, είναι αρχηγός, διευθυντής του γραφείου σας. Συνεχίζει να είναι... Α, είναι μέλος του γραφείου του κύριου Μάλτερ, μάλιστα. Ε, ε συγγνώμη, είναι δηλαδή ακόμα πολύ κοντά μας και θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και τους εισηγητές. Ο Κρίστιαν Ήλερ, εισηγητής. Α, όχι, συγγνώμη. Θα ήθελα να αναφέρω την Τερέζα Μονταρέλ που δεν είναι πια στο Κοινοβούλιο αλλά συμμετέχει ε, στο ορίζον 2020. Τρεις ερωτήσεις έχω. Βρισκόμαστε στην αρχική φάση των διαπραγματεύσεων του ετήσιου προϋπολογισμού ανάμεσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι αναμένετε ότι θα γίνει και ποια είναι η θέση τακτικής της Κομισιόν διότι ανοίξαμε την πόρτα για ένα backloading αλλά ήταν πολιτικός συμβιβασμός ε, και τώρα είναι ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός που θα διαπραγματευτούμε υπό αυτούς τους όρους. Τι περιμένετε λοιπόν όσον αφορά το αποτέλεσμα. Και αυτό σχετίζεται με τη δεύτερη ερώτησή μου. Όσον αφορά τις περικοπές, ε, βρισκόμαστε στη θέση ότι Πιεζόμαστε από δύο πλευρέ. Κάνουμε περικοπέ ε, στο ορίζον, το οποίο οδήγησε σε υπερβολική συμμετοχή σε σχέση με του πόρου. Είχαμε όμως και πολύ έντονη συμμετοχή των κρατών μελών, διότι τα κράτη-μέλη που έκαναν τις περικοπές ε, θέλουν να επωφεληθούν. Συμμετείχα σε μια συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου και είχαν ένα πανό που έλεγε ορίζον ή θάνατος και ε, πρόκειτο για επίσημη διάσκεψη. Οι περικοπές ε, λοιπόν είναι επίσης κάτι που θα σας απασχολήσει και μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για το backloading να δοθεί δηλαδή περισσότερο βάρος σε μεταγενέστερη φάση. Και τρίτον, έχω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις ε, έρευνες και τη συνεργασία στον τομέα αυτών. Ε, είναι το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στις διάφορες περικοπές που θα πρέπει να γίνουν Φαίνεται λοιπόν ότι έχει πέσει θύμα του προϋπολογισμού. Ποιος πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ο ρόλος και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, για τις έρευνες αυτές. Και τρίτον, η ερώτησή μου σχετίζεται με το θέμα της απλοποίησης. Τι προσδοκίες έχετε, θα έχουμε απλοποίηση αλλά θα ανατίθενται όλο και περισσότερο εργασίες στους διάφορους οργανισμούς. Ποιο είναι το γενικότερο σχέδιο. Θα λειτουργήσει καλά κάτι τέτοιο. Το RTD θα λαμβάνει όλο και λιγότερα χρήματα και κάποιος εξωτερικός οργανισμός ε, θα ε, ε, διανέμει τα χρήματα. Ποια θα είναι η δομή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μόντε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή και σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε τη σημασία που δίνουμε εμείς ως Επιτροπή στο πρόγραμμα Horizon 2020. Κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την απλοποίηση που σχετίζονται με την χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Πρώτον, όσον αφορά το κόστος ε, του προσωπικού και αν θα ασχοληθείτε με το θέμα του νέου συστήματος, ε, του ετήσιου υπολογισμού δηλαδή και όχι του μηνιαίου που ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, όσον αφορά την απλοποίηση των, ε, του εσωτερικού κόστους και την δυνατότητα να ε, αναφέρεται το κόστος των προγραμμάτων ε, όχι ως ε, άμεσο κόστος του προϋπολογισμού και κάτι ακόμα. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που πρότεινε ο Επίτροπος Μόιτας στο Συμβούλιο και μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μορφή θα έχουν όλα αυτά και πώς θα σχετίζονται με άλλους οργανισμούς όπως το ERC. Και τέλος, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το να διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός ανάλογα με τα αποτελέσματα σίγουρα είναι ζωτικό μέρος του πώς θέλουμε να προχωρήσει ο προϋπολογισμός. Εξετάζοντας ε, κάποιους από τους στόχους που υπάρχουν ε, στον παρόντα προϋπολογισμό θα έλεγα ότι συχνά είναι θολή οι στόχοι, άλλα πράγματα απουσιάζουν τελείω. Πώς λοιπόν θα ταιριάξουν όλα αυτά με τον προπολογισμό που θα ε, υποβάλλεται με βάση τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από το ECR, ο κύριος Σάνκερ, αντιπρόεδρος μας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα να είναι ανοιχτό και για άλλες χώρες. Έχω μια ερώτηση σχετικά με δύο, μη, ε, με δύο χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία με την Ελβετία και με την Ρωσία σε τι βαθμό εμποδίζεται ή επηρεάζεται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την Ελβετία μετά την ε, ψηφοφορία για τη μετανάστευση και με τη Ρωσία μετά την επιβολή κυρώσεων. Η δεύτερη ερώτηση που έχω σχετίζεται με τη γραφειοκρατία. Αναφέρατε ότι Το 14% των προγραμμάτων εγκρίνονται επιτυχώς. Δηλαδή 14 ε, ενότητες από τις 100 ε, είναι ικανοποιημένες ε, με τις αποφάσεις, οι υπόλοιπες 86 όμως δεν είναι. Με ανησυχεί ο αντίκτυπος στην επιστημονική κοινότητα, διότι υπερβάλλω λίγο, αλλά η προσωπική μου εμπειρία μου δείχνει ότι οι επιστήμονες της Ευρώπης ασχολούνται όλο περισσότερο με την σύνταξη προτάσεων και όλο και λιγότερο με την έρευνα, που νομίζω ότι ήταν ο αρχικός στόχος. Στο πλαίσιο αυτό έχω άλλη μια ερώτηση. Πόσα άτομα απασχολούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση του προγράμματος Horizon 2020, έμεσα και άμεσα, και πώς σχετίζεται αυτό με τον προϋπολογισμό και πώς έχει εξελιχθεί η δομή αυτή κατά τη διάρκεια των τελευταίων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το λειτουργικό κόστος που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε παραμένει στο ίδιο ποσοστό ή αυξάνεται ή μειώνεται. Και μια ερώτηση που έθεσα και στον Επίτροπο Μόεντα την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήθελα όμως να τη θέσω και εσάς. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα πολύ να ε, μου απαντήσετε κάποια στιγμή. Οι ανθρωπιστικέ σπουδές και οι κοινωνικέ επιστήμες θα πρέπει αμέσω να καλύπτονται από το ορίζον 2020 με την ιδέα της ενσωματωμένης έρευνας. Θα ήθελα λοιπόν να έχω αποδείξεις ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Διαβάζοντας ε, το ε, έντυπο αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικό και τα συγχαρητήριά μου γι' αυτό, υπάρχουν παραδείγματα προγραμμάτων, αλλά ούτε σε ένα από αυτά δεν μου δόθηκε η εντύπωση ότι έχει ενσωματωθεί η έρευνα για στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σήμερα στις ερωτήσεις μου, θα ήθελα πολύ να τις λάβω σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας ή ενδεχομένως γραπτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Τεπάκερ από την Άλτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Κάποιες ερωτήσεις από τη δική μου πλευρά. Αναφέρατε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι η υπερβολική συμμετοχή που οφείλεται εν μέρη στην επιτυχία των προγραμμάτων, ε, οφείλεται όμως και στην ε, περικοπή ε, του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και η γενική ποιότητα των προγραμμάτων, είπατε, είναι πιο υψηλή. Ταυτόχρονα αναρωτιέμαι, έχετε αλλάξει κάτι στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, διότι εάν αυτή έχει διατυπωθεί με ευρύτερο τρόπο, τότε πιο πολλές ομάδες μπορεί να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα, αυξάνοντα έτσι και τον αριθμό των αιτήσεων. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα κράτη-μέλη, παρότι λένε πολλά πράγματα για τις έρευνες, και τη σημασία της έρευνας για τις οικονομίες τους. Μέχρι τώρα οι συζητήσεις σε άλλες επιτροπές ε, δεν έχουν λάβει υπόψη τους ότι κάτι τέτοιο θα ε, απαιτήσει περισσότερη χρηματοδότηση και από ε, δημόσιες και από ιδιωτικές πηγές. Σε τι βαθμό λοιπόν τα κράτη-μέλη ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική τους με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Είναι σημαντικό να γίνονται στρατηγικές επιλογές με βάση την ε, καινοτομία που δημιουργείται στα κράτη-μέλη, αλλά μήπως θα πρέπει και η Κομισιόν να αναζητήσει συμμάχους στα κράτη-μέλη, ώστε στον επόμενο γύρο ε, διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό να μπορέσουμε να πετύχουμε επιπλέον χρηματοδότηση για τα προγράμματα αυτά, ιδιαίτερα για την βασική έρευνα. Η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με το κομμάτι του Horizon 2020 που χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και νέες επιχειρήσεις. Εάν δεν υπάρχει μια ευρύτερη προοπτική, θα ξεκινήσουν πολλές μικρές ε, επιχειρήσεις, ε, νέες επιχειρήσεις, μετά από κάνα δύο χρόνια όμως θα διαλυθούν. Πώς λοιπόν σχετίζεται το δικό σας πρόγραμμα με άλλα προγράμματα που να διασφαλίσουν την την ε, χρηματοδότηση ε, και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ε, και τέλος, πολύ συγκεκριμένα για τη γραφειοκρατία. Μήπως πιστεύετε και εδώ ότι τα πανεπιστήμια είναι καλύτερα οπλισμένα ώστε να γνωρίζουν ότι τα προγράμματα που υποβάλλουν συνάδουν με τους στόχους της Κομισιόν και αν όχι τι μπορεί να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τους πράσινους κάποιος. Από την ΚΟΕ όμως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Yeah. Ε, κύριε Σμιτ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ε, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 μπορεί πράγματι να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο για την πρόθεση της έρευνας και της καινοτομίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να προωθήσει την κοινωνική ανάπτυξη. Δυστυχώ όμως, αντί το πρόγραμμα <clears throat> να προωθείται και να δυναμώνεται, δυστυχώ λόγω των περικοπών αποδυναμώνεται συνεχώς. Με την απόφαση δε να δοθούν 2,7 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, οι ελλείψει και οι αδυναμίες που προκύπτουν είναι πολύ σοβαρέ και λειτουργούν βέβαια σε βάρος των συμφερόντων και των αγκών της κοινωνίας. Ε, το πρώτο ερώτημα είναι πώς σκοπεύετε να καλύψετε το μεγάλο κενό πώς σκοπεύετε να καλύψετε το μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση και ποια μέτρα θα προφήσετε ώστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω ακριβώς αυτής της μεγάλης περικοπής. Ιδιαίτερα δε δηλαδή, όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μα είχατε πει κύριε Σμιτ πέρσι τον Νοέμβριο όταν είχατε έρθει ξανά στην επιτροπή μας, πώς μελετάτε διάφορες μεταρρυθμίσεις για απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ένα, ένα χρόνο μετά, ποιε προτάσεις ε, έχετε προωθήσει για να στηρίξετε ακριβώς αυτή την αλλαγή, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, γιατί σήμερα στην εισαγωγή σας δεν ακούσαμε κάτι το συγκεκριμένο. Και το τελευταίο ερώτημα που κλείνω είναι ε, ποια μέτρα θα λάβετε ώστε μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 να επιτευχθεί ένας στόχος που έχουμε θέσει όλοι, δηλαδή τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην άπτυξη νέων προϊόντων, στη μεγέθυνση της οικονομίας και στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κάπελ. Από την ΕΝΕΦ. E ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και μας δείξατε ότι ο Ορίζον 2020 είναι ένα πραγματικό success story, ήταν και στο παρελθόν αλλά και παραμένει και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μας, το είπε και ο κύριος Έλε, να στείλουμε αυτή την επιστολή προς τον κύριο Μοέντες, στον Επίτροπο και να πούμε να μην πάρει τα χρήματα από τον ορίζοντα 2020 ούτε από το Connect Europe για να τα μεταφέρει αλλού. Ήταν σωστή αυτή η κίνηση και καλό το βήμα. Και ρωτώ τώρα τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Την επόμενη περίοδο θα πρέπει να διαπραγματευτείτε. Ορίζον 2020 να έχει τη σωστή πρικοδότηση. Εσείς τι βήματα θα κάνετε από εδώ και πέρα. Και μια ακόμη ερώτηση. Είπατε ότι το 1 τρίτο της παγκόσμιας γνώσης ε, παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο της. Καλά κάνει και δεν θα πρέπει να μειωθεί αλλά να αυξηθεί. Εκεί τι βήματα θα κάνετε και τι ε, βήματα ε, προτίθεστε να κάνετε στη συνεργασία με τρίτες ε, χώρες, τις ανέφερε και ο κύριος Χέγκερ. Εμείς μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρετε ότι σήμερα πολλή γνώση παράγεται σε τρίτε χώρες. Τι κάνουμε με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, με την Νότια Κορέα, πώς συνεργαζόμαστε, μεγάλα θέματα όλα αυτά. Και ένα ακόμα, η συμπερίληψη των επιχειρηματιών και των εμπειρογνωμόνων που έχουν οι επιχειρηματίες το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Το συζητήσαμε και με τον κύριο Μοέντα. Τι έγινε, προχωρήσαμε καθόλου και ποια ε, θα είναι η επόμενη πορεία μας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ερωτήσεις. Εδώ ολοκληρώνει το πρώτος γύρος των ερωτήσεων από πλευρά συντονιστών και αρμοδίων συναδέλφων για το θέμα. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γενικό Διευθυντή να δώσει μία απάντηση. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ ε, τους βουλευτές. Ο κύριος Έλερ αναφέρθηκε ειδικά στον προϋπολογισμό. Αν κοιτάξουμε τις πιστώσεις πληρωμών, συστηματικά είχαμε περικοπές από το Συμβούλιο για τις πληρωμές, επαναλαμβάνω, τις πιστώσεις πληρωμών. Αυτό που οδήγησε, έχουμε σήμερα την κατάσταση, ότι μας λείπουν ένα δις σχεδόν για τις πιστώσεις πληρωμών. Πώς το αντιμετωπίζουμε αναβάλουμε τις προκήρυξεις διαγωνισμών, μειώνουμε τις προκαταβολές, ε, τα βγάζουμε πέρα, τα διαχειριζόμαστε, αλλά κάποια στιγμή αυτό ο λογαριασμό θα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα έργα του 7ου προγράμματο πλαισίου και μόνο που συνεχίζει, που χρειάζονται 9 δι στι πιστώσει πληρωμών ε, για να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον πιστοτική κάρτα χρησιμοποιούμε. Κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμό και λέμε συχνά και συνεχώ στο Συμβούλιο μην κόβεται από εκεί τις πιστώσεις πληρωμών και ευτυχώ το Κοινοβούλιο πολύ συχνά επαναφέρει τις πιστώσεις πληρωμών για το Horizon 2020 και το πρόγραμμα πλαίσιο 7 ε, αλλά αργά ή γρήγορα θα το βρούμε μπροστά μας και θα ε, σκάσει τα χέρια μα Τα διαρθρωτικά ταμεία ε, έχουν κάποιες καθυστερήσεις και σιγά σιγά προχωράνε, αλλά γύρω στο 17-18 θα υπάρχει τεράστια ανάγκη ε, για πληρωμές και για τα διαρθρωτικά ταμεία και ε, για το Horizon 2020 και θα το βρούμε μπροστά μας. Τώρα για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι δύσκολο να αποφανθούμε. Ε, διαβουλεύεται αυτό τον καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Η συνεργατική έρευνα, συμμετοχική, αν έχει υποφέρει, δεν είμαι βέβαιος όλα αυτά τα χρόνια. Αν κοιτάξετε τα μεμονωμένα προγράμματα, το ERC και το Marie Curie δεν είναι η ε, των χρημάτων. Δηλαδή δεν ε, χρηματοδοτούμε κανονικά με μονομένους ερευνητές, μάλλον συνεργασίες. Αν κοιτάξετε τις ΔΙΤ που κάνουμε, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή τη συνεργατική έρευνα, ε, είναι συλλογικές προσπάθειες. Ο κύριος Ελέ ρώτησε και για την απλούστευση, για την απλοποίηση. Το δεν χειριζόμαστε τα προγράμματα και... Ε, χάρη σε αυτούς τους εκτελεστικούς οργανισμούς που δημιουργήσαμε Υπάρχει και κατανομή και επιμονισμός εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάζει τον προγραμματισμό και την πολιτική και ο εκτελεστικός οργανισμός εκάστοτε διαχειρίζεται τους διαγωνισμούς και τις ε, πληρωμές. Αυτά λειτουργούν πάρα πολύ καλά και έχουν οδηγήσει και σε μείωση κόστους. Αν σας πω ότι ένας από τους οργανισμούς για την έρευνα εκτελεστικός ε, του ERC έχει πάνω από 3% ε, πλεόνασμα με εκτάκτους ε, υπαλλήλους, με εμπειρογνώμονες, με βάση τις ανάγκες, γιατί τα περισσότερα χρήματα αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν στην έρευνα και όχι σε διοικητικές δαπάνες. Ε, είναι πολύ ικανοποιημένοι και οι πελάτες, οι συμμετέχοντες δηλαδή, εάν το συγκρίνουμε με προηγούμενα προγράμματα πλαίσια. Βλέπω εδώ τον πρώην Επίτροπο Λεβαντόφσκι Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς στην έρευνα διαχειριστήκαμε τον προϋπολογισμό και πριν από δύο χρόνια το αναφέρατε και στην έκθεση προς το Κοινοβούλιο ότι η δική μας γενική διεύθυνση έχει απορροφήσει κάθε χρόνο 100%. Ούτε δεκάρα τσακιστή σέντ δεν αφήνουμε, ούτε ευρώ. Ε, τα απορροφούμε όλα και δεν είναι πολλές υπηρεσίες που έχουν τέτοιες επιδόσεις να ε, επιδείξουν. Είναι πάρα πολύ καλή η διαχείριση και πιάνει τόπο τα λεφτά. Επίσης, ε, ε, για τον ε, στη ελέγχωση ρωτήσατε και, το προσωπικό και τα λοιπά. Το full cost, στην απλοποίηση θελήσαμε να ξεφύγουμε από το full cost. Αυτό δεν είναι ικανοποίηση τους πάντες όπως γνωρίζετε και πολλά βρετανικά και ιρλανδικά πανεπιστήμια αλλά και άλλοι δεν είναι πάρα πολύ ευτυχείς με την επιλογή που κάναμε αλλά Πρέπει να σας πω ότι ε, τα περισσότερα από τα προβλήματα που είχαμε στον οικονομικό έλεγχο και το λογιστικό ήταν πάντα με εκείνα τα πανεπιστήμια ή ε, τα, τις εταιρείε που ήταν στο full cost. Δηλαδή είχαμε τεράστια συζήτηση ε, ποιο, θα ήταν το έμεσο και το άμεσο κόστος και πώς ελέγχεις το έμεσο κόστος. Ξέρω ότι δυσαριστήσαμε και κόσμο, αλλά αυτό οδήγησε σε μεγάλη απλοποίηση και σε μείωση των σφαλμάτων. Γιατί είμαι τώρα εδώ ενώπιόν σας και συζητούμε για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τα θέματα τα επιστημονικά, αλλά σε λίγες εβδομάδες θα πάω στην κυρία Γκρέσλε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και θα αρχίσει εκεί πέρα για τους οικονομικούς ελέγχους και ε, για τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Οπότε, καταλαβαίνετε πώς έχουν τα πράγματα. Αναφερθήκατε και στο Συμβούλιο Καινοτομία. Τώρα, ε, με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Μοέντας, ε, το σκεφτόμαστε και μας προβληματίζει. Είναι γεγονός ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων του είπε γιατί δεν έχουμε ένα e ένα κέντρο ερευνών για τις νεοφυείς, ε, του τύπου που ήδη έχουμε και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία αυτό το συμβούλιο. Λοιπόν, ε, μας προβληματίζει αυτό, είμαστε στο στάδιο προετοιμασίας και αρχές του έτους θα το εκδώσουμε. Τώρα, ε, ο προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων, αυτό το activity-based budgeting και μεγάλο σεμινάριο οργανώνεται προσεχώς για την έρευνα όμως θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί πολύ, γιατί πολύ συχνά ε, στην έρευνα πολλές φορές και το μηδενικό αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Ας πούμε στην ιατρική έρευνα έχεις πάρει ένα δρόμο και ανακαλύπτεις ότι είναι αδιέξοδο και αυτό αποτέλεσμα είναι γιατί κλείνει ένας διάδρομος και ανοίγεις μια άλλη πόρτα. Δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει το πρόγραμμα. Προσοχή λοιπόν να μην προσπαθούμε στο μέλλον να έχουμε ένα μέτρο απλοποίηση λέγοντας ότι η έρευνα θα πληρώνεται μόνο αν βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά. Δυστυχώς δεν πάει έτσι και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην υπερβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή. Κύριε Χέγκελ, μιλήσατε για την ε, Ελβετία. Ε, πραγματικά έχει παρεμποδιστεί η συνεργασία μετά το δημοψήφισμα που έκανε η ε, Ελβετία. Συμμετέχει μόνο σε ένα πυλώνα ε, και στο ΙΤΕΡ και σε κάποια άλλα μέτρα, αλλά όχι σε όλα, στο πρόγραμμα πλαίσιο ας πούμε. Και αυτό πραγματικά παρεμποδίζει τη συμμετοχή της Ελβετίας. Για τη Ρωσία που ρωτήσατε, τα πάντα αυτή τη στιγμή είναι σε χαμηλό επίπεδο. Γίνεται η συνεργασία, αλλά σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν. Σωστά είπατε ότι οι ερευνητές μας πρέπει να κάνουν έρευνη και έρευνα και να μην γράφουν προτάσεις Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό ε, ε, μιλάμε για ένα ε, στάδιο σε δύο φάσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό. να κάνουν πρώτα ένα δεκασέλιδο ας πούμε στο σχέδιο της πρότασης και μετά σε απότερο στάδιο να είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή αν κάθονται από το διαγωνισμό και τη δημοπρασία οι ίδιοι επιστήμονες να αφιερώνουν τόσο χρόνο για να συντάσσουν προτάσεις και υποψηφιότητες ε, τότε πραγματικά πάει χαμένο ανθρώπινο δυναμικό για να υπάρχει και μετά ε, επιτυχία 12 με 14%. Στη ΣΥΠΑ τι έγινε και έχει ενδιαφέρον αυτό. Πρόσφατα έδειξε ότι 42% επιστήμονας του χρόνου του το αφιερώνει σε εκθέσεις, σε αιτήσει για χρηματοδότηση. Οπότε οι ΗΠΑ δεν είναι καλό παράδειγμα για το πώς θα εξασφαλίζουμε ότι οι επιστήμονες θα κάνουν αυτό που είναι η δουλειά τους, που είναι η έρευνα. Αναφερθήκατε στους υπαλλήλους που συμμετέχουν. Ε, σας είπα για τους εκτελεστικούς οργανισμούς είναι 3% και υπάρχει το γερμανικό DFG που είναι η γερμανική ερευνητική κοινότητα κτλ. Ε, τώρα, στις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές δεν έχουμε ξεχωριστό πρόγραμμα αφοσιωμένο σε αυτό στον ορίζοντα 2000. Για ποιο λόγο? Ότι η θεωρητικές και κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να ε, είναι πλήρως ενσωνατωμένα. Ας πούμε, Αλτσχάιμερ και Άνια, αυτό δεν είναι μόνο ιατρικό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες στην Ευρώπη θα πληγούν από αυτές τις αρρωσίες. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία, πού θα ζουν, ποιο θα τους φροντίζει. Δεν είναι μόνο ιατρικό το θέμα, δηλαδή μέσα σε ένα ιατρικό project έχεις και τα κοινωνικά και τα ευρύτερα, τα ανθρωπιστικά. Ε, τι έγινε με τους πρώτους διαγωνισμούς, είχαν επιτυχία ε, οι προκήρυξεις εν μέρη. Ακόμα ε, αυτά είναι σε σιλό, είναι περιχαρακωμένα και σε στεγανά. Έχεις από τη μια τις θετικές επιστήμες, τις ιατρικές και τις κοινωνικές. 220 εκατομμύρια έχει δοθεί ένα κονδύλι για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Θα πρέπει να σπάσουν αυτά τα στεγανά, να είναι διεπιστημονική η προσέγγιση και αυτό είναι θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Εξακολουθεί όμως να μας ε, προβληματίζει. Κύριε Ντεμπάκερ, έχετε απολύτως δίκιο. Αναλυτική ε, ήταν προηγουμένως η ε, παρουσίαση και τώρα την έχουμε γενικεύσει κάπως και έχουμε περισσότερες προτάσεις και αυτό μας λένε και οι ερευνητές. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μας έχετε βάλει ένα στενό κορσέ, μας έχετε πει τι να ψάξουμε. Μήπως να μας πείτε τι θέλετε να βρούμε, ποια είναι τα γενικά ενδιαφέροντα, ποια είναι η πρόκληση και θα σας πούμε εμείς πώς θα πάμε εκεί. Και εγώ λέω στους ε, ε, ε, ερευνητές και στους καινοτόμους, Ε, έχετε δίκιο, αλλά δεν μειώνεται έτσι ο αριθμό των προτάσεων. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ευθυγράμμιση με τα εθνικά προγράμματα. Ζητήματα όπω έχουν να κάνει. Και μίλησα για το Αλτσχάιμερ και την Άνια. Αλλά η, κρίση τροφίμων επισητιστική, το ενεργειακό, αυτό απαιτεί να ευθυγραμμίσουμε τα εθνικά προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέγεται κοινό προγραμματισμό. Joint programming. Και κάνουμε βήματα. Ε, και μέχρι τα τέλη του έτους θα γίνει στο Λούντ μια μεγάλη διάσκεψη όπου θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη την ευθυγράμμιση των εθνικών προγραμμάτων. Διότι το θεωρώ από τα σημαντικότερα βήματα προόδου αυτό. Να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό και να ε, συντονιστούν, να ευθυγραμμιστούν τα προγράμματα. Αυτό δεν σημαίνει ε, εξειδίκευση να κάνει ένα, ένα και όλο στο άλλο, αλλά με κοινή δράση. Αναφερθήκατε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ε, την αξία ε, των αποτελεσμάτων να μπορούν ε, να τα χρησιμοποιούν οι εταιρείε. Το είπε και ο κύριος Σιλικιώτης αυτό και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή από το FP7 στο ορίζον 2020. Για πρώτη φορά υπάρχει συνέχεια της έρευνας με την καινοτομία. Πιλωτικές γραμμές 5, 6, 7 επίπεδο, δηλαδή τώρα ε, δεν ε, δίνουμε την ευκαιρία να παράγεται γνώση, αλλά και να αναπτύσσεται και ε, να τη χρησιμοποιούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Η απλοποίηση είναι μια διαδικασία διαρκής και μόνιμη, την ανέφερα και θα συνεχίσω να την προωθώ. Κυρία Κάπελ, τελευταίο και πολύ σωστά είπατε ότι πέρα από τα θέματα τα δημοσιονομικά στα οποία πίνδυσα προηγουμένως, είπατε ότι έχει σημασία να βγούμε και προς τις τρίτες χώρες, να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία με τη την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Θα ήθελα να πω εγώ ότι ορίζον 2020 θα πρέπει να είναι το πιο ανοιχτό πρόγραμμα στον κόσμο. Κάνουμε μεγάλη εκστρατεία για να φέρουμε αυτά τα λαμπρά μυαλά Κινέζους και Αμερικανούς να συμμετέχουν στις προσπάθειές μας. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη καμπάνια, μια εκστρατεία στην οποία έχουμε επιδοθεί και στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε αρχίσει ε, μια πολύ ωραία δραστηριότητα που λέγεται Προορισμός Ευρώπη, Destination Europe. Ξέρετε ότι αιώνες ολόκληρους μας παίρναν τα ταλέντα και τα μυαλά. Τώρα το έχουμε αντιστρέψει και λέμε στους Αμερικανούς ελάτε στην Ευρώπη. Έχουμε πρώτη ω προγράμματα, ερευνητικά κέντρα, το Ερευνητικό Συμβούλιο, ελάτε σε εμά, συνεργαστείτε μαζί μας και πολύ καλά τα πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Συντάβα. Κυρία Κουντρίτσικα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Γενική Διευθυντή για την εξαιρετική του εισήγηση. Ήταν σύντομη, πολύ συγκεκριμένη και πολύ ισορροπημένη και απαντήσατε πολύ καλά επίσης στις ερωτήσεις. Θα ήθελα εγώ τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Όταν δημιουργήθηκε το ορίζον 2020, ε, θέλαμε να δημιουργήσουμε δυνατότητες, ευκαιρίες για μια μια ισορροπημένη συμμετοχή των των με επιστημονικά προγράμματα ε, όπου θα περιλαμβάνονταν και οι περιφέρειες εκείνες οι οποίες γνώριζαν η στέρηση. Εμείς στην Πολωνία έχουμε ένα σημείο επαφής και οι πληροφορίες που μας στάνουν μας δείχνουν ότι συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη αναλογικότητας ανάμεσα στα παλαιά κρατημέλη και τα νεότερα και ότι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν μικραίνει, δεν μειώνεται. Έχουμε πάνω από 70.000 αιτήματα από τα παλιά κράτη-μέλη και 372 μόλις εκατομμύρια ε, για τα παλιά κράτη-μέλη ενώ τα περισσότερα δίση πάνε στα 15 κρατημέλη. Ε, έχουμε λοιπόν ε, ορίσει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε στείλει συγκεκριμένη επιστολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληρωμές των προγραμμάτων αυτών στα νέα κατημέλη για ιστορικούς και διαρθρωτικούς λόγους. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά κάποια λύση για το πρόβλημα αυτό και ποιες είναι οι δράσεις που μπορούμε να αναμένουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, οι παρατηρήσεις σας είναι πολύ σημαντικές. Ε, το έχω δει την επιστολή που στείλατε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε κύριε Γενικέ, ε, για τι πληροφορίες σας ήταν πολύ βοηθητικέ. Όπως είπαμε πρόκειται για έναν αγώνα ε, διακοινοβουλευτικό. Είναι, ήταν αναζωογονητική αυτή η προσπάθεια. Να μην δουλεύουμε λοιπόν απομεινωμένα, αλλά να βλέπουμε ότι ο ορίζοντας 2020 έχει ε, επιπτώσεις ολόκληρη την ατζέντα ε, της έρευνας, τόσο στις ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και στις ε, πρακτικές. Ε, και αυτό το είπαμε το είπε και ο Επίτροπος Μοέδας ότι δηλαδή η με πιθανά εθνικά προγράμματα και μάλιστα η σφραγίδα αριστείας έχει κάποιες δυσκολίες ιδιαίτερα στις αγγλόφωνες περιοχές διότι ε, στις περιφέρειες ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται ε, τα διαστοντικά ταμεία σε εθνικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό. Και αυτό είναι πιο προβληματικό. Έλαβα μια απάντηση από τον Επίτροπο και περιμένω απάντηση από την Κορίνα Κρατσού αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε στο γεγονός ότι ανάλογα το κράτο μέλο οι περιστάσεις που ισχύουν είναι διαφορετικές. Επίσης, οι συνάδελφοι μίλησαν για την προστασία της βασικής έρευνας που δεν μπορεί ακόμα να αποδείξει τι δυνατότητέ τη εμπορικό χώρο. Βορειοδυτική Αγγλία, από εκεί προέρχομαι εγώ, από το Μάντσεστερ και να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ κάνει πολλή δουλειά για να απομονώσει το κύτταρο που μπορεί να οδηγήσει σε ε, εμβολιασμό για το έμπολα. Αυτά είναι πράγματα που ε, είναι χρονοβόρα, αλλά που τελικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις όταν έρθει η επιτυχία. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αλλά και ισορροπία όσον αφορά τους εκπροσώπους της Ασιατικής και της Μαύρης Φυλής μέσα σε αυτούς τους ε, ε, ετούντες. Εξακολουθεί να υπάρχει κενό και ποιες συγκεκριμένε ενέργειες θα λάβετε, θα κάνετε ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά και αυτές οι διαφορές. Ευχαριστώ πολύ κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ πολύ. Η Σνάσφο ανέφερε ότι κατά την έναρξη της συζήτησης για τον ορίζοντα 2020 συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις περιφέρειες που ε, δεν έχουν πολύ ανεπτυγμένη έρευνα. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ομαδοποίησης, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν προωθείται με μεγάλο ενθουσιασμό από την Κομισιόν. Ο αριθμός των προγραμμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένος. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί είναι τόσο δύσκολα όλα αυτά και δεύτερον, γιατί έχουν διαρκέσει τόσο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες. Τρίτον, οι περιφέρειες γιατί δεν χρησιμοποιούν τους εταίρους που ήδη γνωρίζουν. Μήπως ε, χρειάζεται κάποια απλοποίηση. Υπήρχε η πολιτική υπόσχεση στήριξης ε, των περιφερειών ε, που υστερούν. Εάν δεν ασχοληθούμε με αυτό θα έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα να σας καλέσω να γίνουν περισσότερες δουλειές για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τον Επίτροπο Μοέτας για την εκδήλωση της προηγούμενης εβδομάδας όπου ήταν παρόν και ο πρόεδρος Μπούσεκ. Είχαμε λοιπόν το πρόγραμμα που θα ενημερώνει περισσότερο τους ευρωβουλευτές σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα το πρόγραμμα αυτό είναι πολιτική προϋπόθεση για να έχουμε περισσότερη έρευνα, επιστημονική έρευνα και χαίρομαι που λειτουργεί καλά. Δεύτερον, έχουμε και το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ να διαθέσουμε περισσότερους πόρους. Ερώτηση λοιπόν μετά τις ε, δια εφόσον συμμετέχω στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό του 2016, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το μέσο και να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις από τον ανταγωνισμό των εισαγωγικών με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, ε, τι γνώμη έχετε για την ιδέα να επικεντρωθούμε στους μετανάστες στα προγράμματα μας, πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Κάποιοι μετανάστες ε, έχουν πολλά προσόντα τα οποία χρειαζόμαστε. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτούς τους επιστήμονες και ερευνητές. Ίσως θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ποσόστοση, διότι όλα τα κράτη-μέλη θα θέλουν αυτούς τους ερευνητές, ε, δεν, μπορεί, δεν μπορούν όμως ε, να πάνε όλοι σε ένα κράτος. Ε, ευχαριστώ κύριε Σαφχάζη. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά, δύο σχόλια. 20 χρόνια Έχω εργαστεί σε ε, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα δεν έχει προβλέψει τίποτα για να κρατήσει τους ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ σκέφτομαι δύο εταιρείε συγκεκριμένα, γιατί είναι από την Αλσατία. Ξέρετε ότι και εγώ είμαι από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στο παρελθόν αρμόδιος για οικονομικά θέματα, μπας εδώ και καιρό, ε, είναι η Alstom και η Alcatel αυτές οι δύο εταιρείε από την Αλσατία. Έχουμε αφέμητο ανταγωνισμό και μπορώ να το αποδείξω. Για την Alstom πρόσφατα γράφτηκε και βιβλίο, ενώ για την Alcatel είναι μια παλαιότερη ιστορία για το πώς προετοιμάστηκαν τα πράγματα, τα ξέρω εγώ από τα μέσα και θα μπορούσατε να ακούσετε και να ελέγξετε παλιούς ηθήνοντες, όπου αποσταθεροποιήσαμε εταιρείε που ήταν ε, πανευρωπαϊκά ηγέτιδες στην Ευρώπη για να τις κάνουμε τελικά εταιρείε και αυτό ισχύει για την αλκατέλ και προσεχώς για την Alstom, οι οποίες θα αποδιαρθρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον αγοραστή για ποιο λόγο στο πρόγραμμά σας δεν έχετε προβλέψει και ένα κλάδο που να ε, αφιερώνεται στην διαφύλαξη, στη διατήρηση και στην υποστήριξη αυτών των εταιριών που είναι ήδη ηγέτες, που είναι ήδη κέντρα αριστείας. Αυτούς θα πρέπει πρώτα να κρατήσουμε και να προστατεύσουμε πριν ετοιμάσουμε τους μελλοντικούς ε, ε, leaders. Δεύτερο, για την έρευνα. Δύο στοιχεία υπάρχουν εδώ υπάρχει η θεωρητική έρευνα και η έρευνα στις εταιρείες. Η θεωρητική πολύ καλή και ωραία είναι 2,84 δις για το κεφάλαιο κινδύνου και για την παραγωγή, τη βιομηχανική των νέων τεχνολογιών, των γενοτόμων. Ωραία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να αυξηθεί αυτό το ποσό αφενός και αφετέρου. Αν το αφήσετε στα αρχαία για το τραπεζόν, τότε θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Και το λέω εξιδίας πύρας. χρειάζεται ε, να γίνετε business angels, δηλαδή οι φύλακες άγγελοι των επιχειρήσεων. Και ε, ενδεχομένω να υποστηρίζετε και τα εθνικά προγράμματα που έχουν φοροαπαλλαγές για όσο κέρδος επανεπενδύεται ε, εκεί ας πούμε, όχι 100.000 ευρώ ή 100 εκατομμύρια για τα φυσικά πρόσωπα φοροαπαλλαγές όπως συμβαίνει στη Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συγγνώμη Πρόεδρε που μακρηγορώ κάπως. Η έρευνα στις επιχειρήσεις. Εσείς εκεί αν κατάλαβα καλά τι προτείνετε και τι προωθείτε. Το σημαντικότερο δεν το έχω καταλάβει. Τι πρόγραμμα χρειάζεται. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ένα ευρωπαϊκό επαναλαμβάνω ή μήπως η εταιρεία από ένα και μοναδικό κράτος μπορεί να είναι δικαιούχος Παράδειγμα. Ναι, συγγνώμη, μακρηγορώ. Ε, μια πρόταση, κλείστε παρακαλώ. τις περισσότερες φορές όταν κάνουμε τρία ή τέσσερις ένα πρόγραμμα δεν είμαστε στο ίδιο ε, αποτέλεσμα, δεν καταλήγουμε στο ίδιο από ότι αν ένας μόνος. Το ρωτήστε το ερευνητικό τμήμα της Airbus και θα σας τα πει αυτά και είμαστε τώρα σε δύο χώρες. Αν θέλουμε να συγκεράσουμε δύο-τρεις νοοτροπίες ε, ε, και τα λοιπά, θα είναι μικρότερο το αποτέλεσμα και η αποτελεσματικότητα και περισσότερο το κόστος. Ευχαριστώ κυρία Λόπεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή για την ε, εισήγησή του και για την παρουσία του απόψε εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω ότι είναι λυπηρό που διατηρούνται ε, οι περικοπές στο πρόγραμμα Horizon 2020 με τη στήριξη ενός τμήματος αυτού του κοινοβουλίου. Ενώ έχει φανεί ότι για πραγματική παραγωγική ανάπτυξη είναι βασική η έρευνα και η καινοτομία. Κατά δεύτερο λόγο, αυτή η αναθεώρηση του ορίζοντα 2020 είναι καλή στιγμή για να αναθεωρήσουμε και τις προτεραιότητές μας, ώστε να επιτύχουμε ακριβώς αυτούς τους στόχους που είχαμε θέσει. Και γι' αυτό θέλω να επιμείνω για την ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στα ερευνητικά κέντρα και στα δημόσια πανεπιστήμια, να αναζητηθούν οι συνεργίες με πολιτικές σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής, ώστε να αποφευχθεί η εστίαση όλη τη τεχνολογική δραστηριότητα σε κάποιε μόνο περιφέρειε. Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι μικρομεσαίες και του συνεταιρισμού ω φορεί απασχόληση και να αποφύγουμε ότι θα εξαρτώνται από μεγάλε μονοπωλιακού ομίλου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να οριστούν συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια στην, στην ε, δημόσια ε, έρευνα, βελτίωση τεχνολογική, βελτίωση των συνθήκων ε, υγεία κτλ. Αλλά επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε τις συνθήκες εργασίας των ε, εργαζομένων στα κατημέλια που δυστυχώς δεν είναι οι καλύτερες ε, σε όλα τα κατημέλια ώστε να μπορέσουν σωστά να φέρουν σε πέρα στο ερευνητικό τους έργο και τη δουλειά τους γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλήτρια ήσασταν. Ε, να συμπληρώσω και εγώ μια σύντομη ερώτηση για τον τρόπο συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο του Horizon 2020. Πώς το βλέπετε ανάμεσα σε, στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Έρευνας και, τεχνο, και Τεχνολογίας και Καινοτομίας, υπό την εποπτεία δηλαδή διαφορετικού επιτρόπου ναι. και ναι. τους υπόλοιπους τα υπόλοιπα προγράμματα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ε, μέσα στο πλαίσιο του Horizon 2020. Σας ευχαριστώ. Επειδή εσείς είστε το αφεντικό, ξεκινάω απαντώντας σε εσά. Η συνεργασία εντός της ε, Κομισιόν με τους συναδέλφους είναι πρώτης τάξεως. Ε, επειδή το Ερευνητικό Συμβούλιο και το Ερευνητικό Κέντρο είναι τοποθετημένα εκτός της Κομισιόν, χρειάζεται τακτική επαφή για να συζητάμε την πρόοδο το κέντρο για να δούμε πώς οι κοινότητες γνώσης, οι μπορούν να ε, έχουν επαφή, πώς θα εντοχθούν αυτές στα δημοσιονομικά μας μέσα. Ε, η συνεργασία λοιπόν γίνεται πολύ αγαστά και σε επίπεδο γενικών ηθιντών όσο και σε επίπεδο επιτρόπων. Για να έρθω τώρα στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Η κυρία Προντζίσκα μίλησε για το θέμα ο ρήγματος που υπάρχει ανάμεσα στα παλιά, ε, παλιές χώρες και τις νέες χώρες μέλη της Ένωσης. EU15, EU28. Ε, ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω κανέναν λόγο να πανικοβληθώ γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή πιστεύω δεν είναι τόσο επιδεινωμένη σε σχέση με το, πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση. Οι στατιστικέ και τα στοιχεία για τη συμμετοχή ε, παίρνουν τελείως άλλο νόημα όταν διορθωθούν. Αν δούμε σε απόλυτους όρου. πού πάνε τα λεφτά, Βεβαίω βλέπει ότι οι μεγαλύτερε χώρε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, παίρνουν τα περισσότερα χρήματα. Αν όμω το διορθώσουμε και δούμε ποιε είναι οι δαπάνε σε εθνικό επίπεδο στην έρευνα ή τον αριθμό των ερευνών σε εθνικό επίπεδο, βλέπετε μια τελείω διαφορετική εικόνα. Με άλλα λόγια, αν μια χώρα δαπανά μόνο, μόνο 0,1% του εθνικού της προπολογισμού στην έρευνα, δεν είναι εντυπωσιακό που αυτή η χώρα δεν μπορεί να συμμετέχει πολύ καλά στο ορίζον 2020, διότι δεν έχει την επιστημονική βάση. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όταν βλέπουμε τα στοιχεία και ερμηνεύουμε με βάση αυτά τη συμμετοχή. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ πολύ στενά. Τώρα, διάδοση της αριστείας και διεύρυνση των συμμετεχόντων. Και εσείς φύγρατε το πρόγραμμα Teaming. Θυμάμαι τη συζήτηση στη Λάρνακα στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Ήταν δική σας εφεύρεση και είναι ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενο, ε, υποσχόμενο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αναφέρατε λοιπόν το teaming και είπατε ότι είχατε την εντύπωση πως δεν το ε, ε, υποστηρίζει η Κομισιόν ένθερμα. Ε, αντίθετα σας διαβεβαιώ κύριε Ρόιλ ότι έχουν διοργανωθεί δύο συνεδριάσεις στην Πολωνία, στη Βαρσοβία γιατί ακριβώς η ομορφιά της πρωτοβουλίας teaming ε, Ομαδοποίηση είναι ακριβώς στην πράξη η συνεργασία ανάμεσα στον ορίζοντα 2000 και το 2020 και το διασωτικά ταμεία. Είναι οι προτάσεις που επιλέγονται από εμά, ας πούμε, ε, ας πούμε για μια, ε, μια συνεργασία ανάμεσα σε κάποιο βουλγαρικό και κάποιο πολωνικό κέντρο μέσω των οποίων φτιάχνουμε νέα, νέους θεσμούς η πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθεί από το Horizon 2020, αλλά τελικά θέλουμε οι ίδιες οι περιφέρειες να μπορέσουν να επενδύσουν σε αυτά τα κοινά προγράμματα, γιατί αυτό δείχνει τη δέσμευση των περιφερειών μέσω των διαρθωτικών ταμείων να επενδύσουν σε αυτά και να σημάνουν την αλλαγή. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι, θέλουν πολλοί να δουν τις επιτυχίες, επιτυχία και πολλές χώρες μας λένε αυτή είναι η μεταρρύθμιση που θέλουμε. Να έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους προγράμματα και θέλουμε να δώσουμε χρήματα εκεί. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα κύριε Ρόιλ αν μπορούσατε να συμμετέχετε σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις που έχουμε ε, σε υψηλό επίπεδο για να συζητήσουμε την πρόοδο διότι όλοι και η κυρία Κοντρίτσα μπορεί να το επιβεβαιώσει είναι εξαιρετικά ενθουσιώδης για τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, εκτελούνται τα προγράμματα και πώς γίνεται η διαχείριση. Η κυρία Γκοντρίτσκα μίλησε και για το θέμα της αμοιβή, αμοιβήτος μισθούς. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη συζήτηση ε, για τα, από τα 30 ε, κράτη για τους μισθούς. Για τα 13 κράτη που συζητούμε και οι υπουργοί αυτών των χωρών θέλουν να δούμε μήπως μπορούμε να πληρώσουμε υψηλότερους μισθούς ή άλλου είδους μισθούς για, το, ναι. για, για την, τις ε, χώρες της Ευρώπης 13. Κάνουμε λοιπόν μια έρευνα, μια έρευνα στην Πολωνία και μια γερμανική έρευνα στην Βρετανία για να δούμε τους μέσους όρους. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι το κόστος μονάδας για να συζητήσουμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς. Αν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση όμως θα χρειαστεί μεταρρύθμιση των κανόνων συμμετοχής και τότε βεβαίως η δική σας Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα συμμετέχετε ε, πλήρως γιατί είναι μια ε, τέτοια διαδικασία ε, Τώρα, εσείς κυρία Γκρίφιν, σωστά μιλήσατε για προσοχή όταν, σημαίνει, όταν μιλάμε για συνεργασία, συνέργεια και τα διαφορετικά, τις ιδιαιτερότητες των χωρών. Έχετε δίκιο ότι ούτε μία χώρα η περιφέρεια δεν έχει το μονοπόλιο της αριστείας, υπάρχει παντού και πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διάδοση αυτής της αριστείας. Αναφέρατε το παράδειγμα του Μάντσεστερ, όπου τα πράγματα πρώτης τάξης γίνονται ε, εκεί, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Τα περισσότερες επιτυχίες ε, στην ιστορία έχουν προέλθει από τη βασική έρευνα. Αν εστιάζαμε μόνο στην εφαρμοσμένη έρευνα, μάλλον σήμερα θα είχαμε πολύ γρήγορα άλογα, αλλά δεν θα είχαμε εφεύρει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτή η βασική θεμελιώδης έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Ξέρω το πρόγραμμα Γκρίφιν και άλλα προγράμματα τα οποία βασίζονται στην ε, θεμελιώδη έρευνα και γι' αυτό και θέλουμε να συνεργαστούμε το ΣΕΡΝ και που είδατε τι έχει καταφέρει το, τα σκάνερ, ένα σωρό άλλα μηχανήματα ε, που προήλθαν από την θεμελιώδη έρευνα. Ισορροπία τώρα των φύλων. Πολύ μεγάλη προτεραιότητα όντω για τον Επίτροπο Μάδα και για μένα. Έχουμε θεσπίσει τον στόχο 40% για τι συμβουλευτικέ ομάδε, αλλά ε, ξεπλήξαμε του πάντε, ε, βάλαμε 50% το, στο 50% το στόχο μα και δείξαμε ότι είναι δυνατόν. Και επίση, σε σχέση με τα ερευνητικά μα προγράμματα, η έρευνα που χρηματοδοτούμε δεν θα πρέπει ποτέ να βασίζεται στο φύλλο. Δηλαδή, αν κάνει κανεί ιατρική έρευνα ή κλινικέ δοκιμέ, θα πρέπει πάντοτε να δει αν είναι ε, η έρευνα πάνω σε άντρε ή γυναίκε. Αν κάνουμε έρευνα γιατί ε, αυτοκίνητα, ας πούμε, ε, όταν κάνουμε δοκιμές θα πρέπει οι κούκλες να είναι και άντρες και γυναίκες στις δοκιμές, όχι μόνο ε, άντρες. Γι' αυτό και, και στα προγράμματά μας βάζουμε και, από τα, και από δύο φύλλα και φροντίζουμε να υπάρχει ισορροπία. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε σε μια από τις επόμενες μας συνεδριάσεις, ώστε να δείτε ότι είμαστε πολύ προσιλωμένοι σε αυτό το θέμα. Κύριε Ρούμπη, μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη πριν μπείτε στην αίθουσα εγώ μίλησα για τη μεγάλη σας συμβολή, συμβολή στην συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Horizon 2020. Αν χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, εδώ δεν βρίσκομαι για αυτό το λόγο. Εδώ, αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία που βλέπετε και η επιτυχία που έχουμε μιλούν από μόνα του. Έχουμε τόσε πολλέ προτάσει που δεν μπορούμε να τι χρηματοδοτήσουμε ε, και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό για του ετούντε που έχουν ε, ε, φιέστατε ιδέε. λαμπρές ιδέε και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα το μεταναστευτικό. Συντάσσουμε μια σχετική έκθεση. Τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά, από το Horizon 2020 και ο ο Πίτροπος το σκέφτεται και ιδιαίτερα όσον αφορά τι θεωρήσεις ώστε οι ε, ε, λαμπροί ε, επιστήμονες να μπορέσουν αμέσως να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια σας. Αυτό είναι το πιο άμεσο και προφανές ε, προφανή βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, ορίζον 2020 δεν είμαστε βιομηχανικό πρόγραμμα, δεν είμαστε πρόγραμμα βιομηχανική πολιτική. Είμαστε ένα πρόγραμμα που αφορά την ε, καινοτομία και την έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εμεί για την Alstom και την Alcatel. Ε, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Εμείς, σύμφωνα με αυτό που ισχύει, δεν είμαστε πρόγραμμα βιομηχανικής πολιτικής και λέμε, ας πούμε, ότι αυτέ είναι εταιρείε που δυνητικά είναι οι νικητές και γι' αυτό θα επενδύσουμε μαζί τους. Ε, δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, απλά λέω ότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της ε, σημερινής πολιτικής, της ισχύουσας πολιτικής. Πρέπει να μιλήσουμε με τα κεφάλαια τα επισφαλή, με τους επενδυτικούς αγγέλους ε, και ε, Όντω, όλα αυτά σχετίζονται με την ιδέα του, του Επιτρόπου Μοέδας, δηλαδή ένα ερευνητικό συμβούλιο για τις μεμονωμένες νεοφυείς startups εταιρείες, αλλά αυτό το μελετάμε στις, στις, ε, στις σκέψεις μας. Κυρία σε συνεργασία με τα διευθυντικά ταμεία, όντως για να υπάρξει μεγαλύτερη επιτυχία και τώρα οι συνθήκε εργασία για του ερευνητέ μέσα στο πλαίσιο της του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα είναι μεγάλη προτεραιότητα. Ξέρετε ότι την αποδείξαμε χάρτη για του ερευνητέ και με χαρά βλέπουμε ότι πολλά πανεπιστήμια έχουν συνυπογράψει αυτό το χάρτη και υπόσχονται και δεσμεύονται για καλέ ε, συνθήκε εργασία για του ερευνητέ. Τέλο, ήταν η δική σα ερώτηση, στην οποία ήδη απάντησα. Έκανα τη δουλειά μου δηλαδή. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά. Έχουμε περάσει κατά 20 λεπτά το χρόνο μας, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενική Διευθυντά που ήρθατε σήμερα μαζί μας και που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Χαίρετε. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 5. Διαφάνεια και σύγκληση στη φορολογική πολιτική στην Ένωση. Η συγκητής μας ο κύριος Μασιμιλιάνος Σαλίνη. Συνάδελφε, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε για πέντε λεπτά το σχέδιο χρηματοδότησής σας. Ε, είμαστε 27 λεπτά πίσω από το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ λοιπόν να μην ξεπεράσετε το χρόνο σας. Συνάδελφε Σαλίνη. La, allora, l'opinion è stata costruita nel tentativo di evitare η γνωμοδότηση συντάχθηκε με στόχο να απευθυνθεί αυτό το θέμα, αυτό το θέμα της ε, φορολογικής, του φορολογικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων να μετατραπεί σε έναν πόλεμο ε, ομάδων ε, ε, Όπω γνωρίζετε, στόχο μα είναι ένα ευρωπαϊκό. Ε, μάλλον έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τα φορολογικά συστήματα είναι πολύ διαφορετικά στις διάφορες, ε, στα διάφορα κατημέλη και στην Ιταλία συγκεκριμένα έχουμε πολύ ψηλότερη φορολογία από ό,τι αλλού. Τα βασικά στοιχεία των οποίων στηριχτήκαμε είναι κυρίω το πακέτο για την φορολογική διαφάνεια τη 18 η Μαρτίου και το πρόγραμμα δράση τη 17 η Ιουνίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντάξαμε λοιπόν μια γνωμοδότηση που στόχο έχει να αποφύγει η έλλειψη ισορροπίας στη φορολογική πολιτική κάθε χώρας ε, να διαβρώνουν ε, την ε, κατάσταση. Δηλαδή ή να υπάρχει διάβρωση ή να υπάρχει λιγοστή διαφάνεια, το πράγμα το οποίο ζημιώνει καταρχήν τις δυνατότητες των επιχειρήσεών μας να λειτουργούν σε περισσότερες χώρες και κυρίως κάνουν πολλές μη ευρωπαϊκές χώρες να φεύγουν τρέχοντας και οι μη ευρωπαίοι επενδυτές πολύ δύσκολα εμπιστεύονται το ευρωπαϊκό σύστημα. Η βασική υπόθεση είναι ότι η φορολογική, ο φορολογικός ανταγωνισμός, αν γίνεται με διαφάνεια, μπορεί να είναι ένα μέσο υπέρ της ανάπτυξης ε, και όχι αντίφαση του ίδιου του συστήματος. Ε, γιατί όπως έλεγα καταρχήν, οι δικές μας επιχειρήσεις σχεδόν στο σύνολό τους λειτουργούν, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να βοηθηθούν να το κάνουν και να μην αποθαρρύνονται. Επιπλέον υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα μάλλον δύο εμβαθύνσεις που θα επέτρεπαν ε, να λειτουργήσουν σαν παραδείγματα. Το πρώτο στο σημείο 5 αναφέρεται στην, στο μεγάλο πρόβλημα της διπλής εφορολόγησης. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει απόλυτα το CCTB, η Κοινή Ενωπημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών, αλλά θέλουμε να υπάρξει και κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές, ώστε ε, τα οι φόροι που οφείλονται σε μια χώρα και έχουν καταβληθεί εκεί να μπορούν να είναι απαλλάξιμα στην χώρα της εταιρείας. Ε, να μην υπάρχει δηλαδή διπλή ε, φορολόγηση, να εκπίπτουν. Έπειτα, ε, έχουν υπάρξει διαφορετικά υποθέσεις ε, για να προτείνουμε την επιλογή συγκεκριμένων περιφερειών που είναι πίσω ή, ή ζώνες νεκρές όπου υπάρχει όπου υπάρχουν μεγάλες φοροαπαλλαγές ή ε, πιστώσεις φορολογικές που να εκπίπτουν στη συγκεκριμένη πρόταση του σημείου 6, δηλαδή ε, παρακολούθηση από πλευρά τη επιτροπή, εδώ εμεί προτείνουμε, να δημιουργηθούν λοιπόν τέτοιων ελευθέρων ζωνών, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση είτε συγκεκριμένων περιοχών, είτε συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητα ε, και ανάπτυξη. Αυτέ είναι βασικά οι προτάσει μα και αν θέλετε φυσικά είμαι στη διάθεσή σα για να αποσαφηνίσω περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε για τις παρατηρήσεις σας πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Την ε, πολιτική για την φορολογία των εταιριών στην Ένωση, επίτευξη διαφάνεια, συντονισμός και σύγκληση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, πρώτα στον κύριο Γιάννη Σκάγερ από το SND. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με τον εισηγητή συμφωνούμε σε κάποια πράγματα και διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι λείπουν από την γνωμοδότηση κάποιες σαφείς δηλώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν από πλευράς της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και πιστεύω ότι στο σημείο 2 θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις όταν διαπιστώνονται επιθετικές πολιτικές φορολογικού σχεδιασμού, φοροαποφυγής, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική διαδικασία και όχι η βάρος των εταιριών που δεν έχουν τα χρήματα να προσλάβουν φοροτεχνικούς που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Η διαφάνεια λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την καταβολή των φόρων. Θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις αναχώρα, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα σημείο για την ψηφιοποίηση και κατά πόσο μπορεί να υπονομεύσει τις εθνικές φορολογικές πολιτικές. Όσον αφορά το σημείο 6, διαφωνούμε με τον εισηγητή. Σπάνια έχει τύχει να διαβάσω έκθεση που να είναι τόσο υπέρ των ε, ζωνών των ελεύθερων ζωνών της Ένωσης. Προσπαθούμε να κλείσουμε τα παραθυράκια φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να εξαλείψουμε τα ευνοϊκά καθεστώτα που δημιουργούνται από τις ανισότητες, ε, από τις διαφορές ε, στη φορολογική πολιτική των χωρών. Το ότι θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τις ελεύθερες ζώνες πιστεύω ότι είναι τελείως λάθος ε, πολιτική. Χρειαζόμαστε λιγότερους φορολογικούς παραδείσους και όχι περισσότερους. Τα φορολογικά θέματα είναι εθνικά θέματα, αλλά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ε, Επίτροπος ε, θα ήθελα να εξαλείψω τις διαφορές. Ε, έχουμε ζητήσει λοιπόν την διαγραφή του σημείου αυτού. Εάν παραμείνει όμως θα πρέπει να καταψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Σαλίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μαραγκάλ. Ξερώμα του Πρασίνων, μάλλον, ε. ε, ε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ακούσω τα όσα είπε ο κύριος Σαλίνη, γιατί ήμουν στην Επιτροπή Πολιτισμού σε άλλη συζήτηση. Αλλά επειδή έχουμε ανταλλάξει απόψει για τη γνωμοδότηση αυτή, πώς να το πω, Έχουμε συναντήληψη. Ε, η έκθεση είναι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και εμείς κάνουμε γνωμοδότηση εδώ και το συζητάει και η τάξη, η Ειδική Επιτροπή. Δηλαδή είναι εγγυημένη πολύ καλή κάλυψη των θεμάτων αυτών που άπτονται των μεγάλων ομήλων και της, ε, των πρακτικών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής για να μεταφέρουν τα κέρδη εκεί και να αριστεύουν ε, στην βελτιστοποίηση τη λεγόμενη, τη φορολογική. Γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ στην Ήτρε η δική μας δουλειά θα πρέπει να είναι διαφορετική. Να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να προσθέσουμε ε, πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δική μας δουλειά. Έρευνα, ανάπτυξη, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια. Ε, αυτή είναι η δική μας αρμοδιότητα, έτσι. Θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όχι μόνο το, το φορολογικό dumping ε, μεταξύ κρατών, αλλά και πώς θα εξασφαλίσουμε ε, την ισορροπία ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους και τον τεράστιο και απέραντο κόσμο των μικρομεσαίων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν ξέρουν αυτά τα μοντέλα, αυτό ε, το νεφέλωμα Και ο κοινό παρονομαστής είναι ε, η μειονεκτική τους θέση. Δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα τη διαπραγματευτική, ούτε τα μέσα που έχουν οι μεγάλοι όμιλοι στη διάθεσή τους που χρησιμοποιούν και πολλές φορές, καμιά φορά χρόνια κιόλα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ουσιαστικό φορολογικό και αποτελεσματικό φορολογικό συνδελεστή, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ. 30% είναι θεωρητικά στην Ισπανία η φορολογήση των επιχειρήσεων, αλλά μεγάλη όμιλη είναι 5-6% ουσιαστικά. Άλλη ανισορροπία που θα πρέπει να σπάσει είναι να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική οικονομία, την καινοτόμα που παράγει ε, και στην κερδοσκοπική, την οικονομική και την οικοδομική που δεν ε, προσφέρει στην πραγματική οικονομική ζωή. Επίσης, θα πρέπει να προωθηθούν οι επενδύσεις στο κοινωνικό κεφάλαιο, τα equity δηλαδή, ε, τις ιδιωτικές μετοχές, για να ε, αντισταθμιστεί η σημερινή κατάσταση που ευνοεί ε, τη χρηματοδότηση μέσω της, ε, της έκδοσης δημοσίου χρέους που συνοδεύονται από φορολογικά κίνητρα και ευνοϊκή μεταχείριση. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται με την κατάρτιση, την γενοτομία και την έρευνα και την έρευνα, ε, την, ε, την ελεύθερη έρευνα, την απρόσκοπτη και μάλιστα εκείνη που δεν συνοδεύεται από διπλώματα εύρεση τεχνίας. Υπάρχουν έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή απόδοση κτλ. Ε, τέλος, εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο CCC, την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών, με τρία όχι με δύο, για να υπάρχουν πραγματικές ενότητες φορολογικές ευρωπαϊκές. Και συμφωνούμε να τεθεί αμέσως σε ισχύ το συντομότερο της έκθεσης αναχώρα, αυτό το country by country, είναι μια σωστή και λογική ε, πρόταση του κυρίου Γιούνκερ. Δηλαδή να φορολογείται κανείς εκεί που παράγει το κέρδος. Αυτά όλα μας ενδιαφέρουν και όχι περιπτωσιολογία γιατί πολύ συχνά η ε, υπερβολική ρύθμιση παράγει τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα εργαλείο που μπορεί να είναι κίνητρο και ενθάρρυνση, όπως είναι φορολόγητες ε, ζώνες, οι ελεύθερες ζώνες αυτές tax free, δεν θα πρέπει να γίνουν αυτοκινητόδρομοι προς νέους παράνομους φορολογικούς παραδείσους. Ελπίζω και είμαι βέβαιος, όχι ελπίζω, ότι θα προχωρήσουμε και θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάλλος από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη που άργησα. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να είναι απλό το φορολογικό σύστημα. Στην Εστονία δεν έχουμε φοροτεχνικούς, έχουν χάσει τη δουλειά τους επειδή είναι τόσο απλό το σύστημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο σημείο 6 που αναφέρεται η θέσπιση προσωρινού προγράμματος ελεύθερων ζωνών της Ένωσης, αναφέρεται στις ε, φορολογικές παρεκκλήσεις, στις φορολογικές εκτόσεις. Εάν υπάρχουν αυτές όμως, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιστοποιήσει κανείς ε, τους φόρους, να βρει τους καλύτερους φοροτεχνικούς, ώστε να δικαιούται διάφορες φορολογικές εκτόσεις και έτσι δεν πληρώνουν όλοι το δίκαιο μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν τους καλύτερους φοροτεχνικούς και νομικούς. Και μπορούν έτσι να βελτιστοποιήσουν την, την καταβολή των φόρων, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν από κάτι τέτοιο. Ε, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. για την πρότασή σας, της απλοποίησης δηλαδή. Η κυρία Κάπελ από το ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια, ήθελε όμως να πω λίγα λόγια για την έκθεση αυτή, διότι είμαι μέλος ε, και της ε, ΕΚΟΝ ε, και της ΤΑΞ και θα ήθελα να πω ότι Γενικά βρίσκω πετυχημένη την έκθεση αυτή του συναδέλφου Σαλίνη. Μπορώ να συμφωνήσω με τα περισσότερα από όσα λέω. Πιστεύω ότι είναι καινοτόμα η πρότασή του στο σημείο 6. Όσον αφορά την ε, κοινή φορολογική βάση, να μην κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι με κάτι τέτοιο δεν θα υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη. Ε, θα υπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει. Η φορολογική βάση όμως θα πρέπει να είναι ενιαία ώστε να μην έχουμε φοροαποφυγή και επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Όσον αφορά τα σημεία 4 και 5 που αναφέρθηκαν, ε, που αναφέρονται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ε, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ε, είναι πολύ σημαντικά. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα μέσα της επόμενης χρονιάς. Τον Οκτώβριο περιμένουμε από το Συμβούλιο σχετική γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι η έκθεση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφωνίες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από ε, την Κομισιόν όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ε, φορολογικές αποφάσεις. Ε, το θέμα λοιπόν είναι ποιοι θα έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό μεταξύ αυτών των τριών εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την έκθεση Σαλίνη, την έκθεση Φέρβερ και το σχέδιο που ε, συζητάμε, την ε, Φερέρα Τόιρε. Θα πρέπει να υπάρχει ε, συνάφεια μεταξύ αυτών των τριών εκθέσεων, διότι αν δεν υπάρχει, επιδεινώνουμε τη θέση μας απέναντι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεννόηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας αυτές. Η κυρία Λόπες. Συγγνώμη που άλλαξα τη σειρά των ομιλητών. On behalf of ναι. uh, GUE, of course. No hay ningún problema, Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι... Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικό από τώρα να γίνει συντονισμός στην φορολόγηση των εταιριών και είναι σημαντικό κυρίως για την βιομηχανία γιατί είναι σημαντικό να αποφευθούν οι καταστάσεις όπως το φορολογικό dumping γιατί έτσι δημιουργείται ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω πλευρά των ε, βιομηχανιών, πράγμα το οποίο δημιουργεί και πίεση κατά συνέπεια στις ε, μισθολογικέ ε, καταστάσεις που επικρατούν στις χώρες, αλλά και στα πόσα κονδύλια υπάρχουν για επενδύσεις. Οι μέτοχοι απαιτούν ε, μερίσματα, αυτά που όσο γίνεται μεγαλύτερα και όσο γίνεται μικρότερη φυρολόγηση για τις εταιρείες του. Σημαίνει επίσης απώλεια κερδών για την ε, επιχείρηση, για την εφορία, που σημαίνει με τη σειρά του με λιγότερες δημόσιες επενδύσεις και αδυναμία ανάκαμψης. Θέλουμε η φορολογία να χρησιμοποιείται για θεμητούς λόγους, όπως η ανάπτυξη της απασχόλησης και της τεχνολογίας, της τεχνολογικής έρευνας σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Θέλω να τονίσω ότι είναι παράξενο που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αφιερώνει τόσο πολύ χρόνο να ερευνά για δημόσιες ενισχύσεις ή να φορολογεί εταιρείε οι οποίες είναι παραγωγικές και δίκαιες κοινωνικά, ενώ όσον αφορά τα tax ruling, τα ειδικά ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα, να μην ασχολείται τόσο πολύ, ε, ούτε καν ε, ε, όσο θα έπρεπε μετά από το σκάνδαλο του Λίξ. Τέλος, για τις ελεύθερες ζώνες. Ε, μας ανησυχεί αυτή η πρόταση, γιατί θα ήταν κάτι που θα οδηγούσε σε μια κατάσταση φορολογικού παράδεισου. Άνευ φόρων δηλαδή θα ήταν αυτές οι ζώνες και εδώ είμαστε αντίθετοι. Είναι η κόκκινη γραμμή για μας. Αντίθετα θα πρέπει να υπάρξει κάποια φορολογική, ένας βαθμός φορολογικής εναρμόνισης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, να συγχαρώ τον συνάδελφο Σαλίνη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες καλά πληρωμένες ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένας αγώνας ε, αναδιανομής από τη μία ε, όσον αφορά την φορολογία και από την άλλη όσον αφορά ε, τα κέρδη των επιχειρήσεων που να μπορούν να επενδύσουν. Θέλουμε λοιπόν τα χρήματα να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα ε, στους ε, εργοδότες να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ε, μόνο κάτι που έχει παραχθεί μπορεί να διανεμηθεί και αυτό ουσιαστικά είναι το αποφασιστικό. Φυσικά μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν βελτιστοποιήσει τον τρόπο καταβολής των φόρων τους το 4 Ε, τα 100 των φόρων πληρώνουν ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, και το 18 πληρώνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. αν όλοι πληρώνουν το ίδιο, τότε θα είναι πιο ευνοϊκό το καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. θα πρέπει λοιπόν η κατανομή να γίνει με τρόπο ουδέτερο, ώστε να υπάρχουν χρήματα για ε, επενδύσεις και έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό και στις περιοχές όπου είναι μεγαλύτερη η ανεργία θα πρέπει να ε, σκεφτούμε με τρόπο καινοτόμο πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, πώς μπορούμε να τους δώσουμε μία ανάσα ώστε να καλύψουν το κόστος ίδρυσης. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα της εταιρική φορολογίας ώστε να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις. Έτσι θα μπορέσουν να δημιουργηθούν καλές θέσεις απασχόλησης και να γίνει και σωστή η εισπραξή των φόρων. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον συνάδελφο Σαλίνη διότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά αυτή που θα ε, θέσει την Ευρώπη σε νέα θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Γενική Διεύθυνση Ταξούντ, ο κύριος Ήρη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να σχολιάσω τα όσα υπόθηκαν. Καταρχάς είμαστε ευγνώμονες για την επικοδομητική προσέγγιση τα σημεία 1 3 απόλυτα με την πολιτική της Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο σχέδιο δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει υποχρεωτική την ε, κοινή ενωπημένη φορολογική βάση για τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν φορολογικές ευκαιρίες για τις ε, πολυεθνικές εταιρείες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να ε, έχουν ε, την, να εκμεταλλευτούν τις ίδιες ευκαιρίες. ότι η, η Υπουργοί Οικονομικών ε, θα βρουν μια λύση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και σχετικά με την αυτόματη αλλαγή πληροφοριών ε, για τις ε, φορολογικές αποφάσεις. Όσον αφορά τις φορολογικές πιστώσεις, αυτό είναι ένα σημείο που συνάδει με τις συστάσεις μας του 2009 σχετικά με την βελτίωση της ε, πιο γρήγορης καταβολής των πιστώσεων. Στηρίζουμε λοιπόν και επικροτούμε τον τρόπο που ο κύριος Σαλίνη έχει διατυπώσει το σημείο αυτό. Στο σημείο 6 θα ήθελα να είμαι πιο επιφυλακτικός διότι αυτό το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων των συναδέρφων στην ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ε, κάθε θέμα ε, ελεύθερων ζωνών στην Ένωση άπτεται των θεμάτων κρατικής ενίσχυσης. Έχουμε για παράδειγμα την Μαδέρα. Υπό κάποιες προϋποθέσεις μόνο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που προτείνει ο συνάδελφος Αλήνης στην παράγραφο 6. Αυτά είχα να πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Πρόεδρες, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της και θα ήθελα να δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή, διότι ακούσαμε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι δεν συμφωνούν όλοι με το σύνολο της πρότασής σας. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις τελικές σας παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι παρατηρώ ότι υπάρχει μια γενικά θετική διάθεση σχεδόν για το σύνολο αυτή τη γνωμοδοτησή μου. Μια μικρή πρόκληση, γιατί και μεταξύ μα ε, ε, καλό είναι που και που να μιλάμε και για καθόδη πράγματα για να ξεφάγουμε και από την ανία. Mm που πολλές φορές ε, μας ε, ε, ταλανίζει και να μπορέσουμε να δουλέψουμε για κάποια πράγματα τα οποία να έχουν στόχο τις αλλαγές. Το θέμα των ελευθέρων ζωνών που είναι νομίζω το μόνο το οποίο αναφέρθη ως περίπλοκο κατά τη δική μου προσωπική, από τη δική μου μάλλον προσωπική εμπειρία τόσο από πολιτική άποψη όσο και από επιχειρησιακή άποψη είναι ένα μέσο το οποίο είναι το εντελώ αντίθετο του ε, φορολογικού παραδείσου γιατί οι ελεύθερε αυτέ ζώνε. Ε, ε, τι, τι, τι εμπειρία υπάρχει όσον αφορά στην Ευρώπη και σίγουρα και στην Ιταλία. Ελεύθερες ζώνες γίνονται εκεί όπου υπάρχουν μικρές ε, ε, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση. Είναι το μέσο ώστε η αγορά να βοηθηθεί να ανακάμψει και είναι ένα μέσο που κανονικά ελέγχεται από το κράτος, ώστε ούτω ώστε να μην γίνουν ο νόμος ή ο κανόνας και να δημιουργήσουν ε, αδιαφάνεια και έλλειψη ισορροπίας με άλλες καταστάσεις. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται ως μέσα ισότητας με χρυσό του μια διαφορετική κατάσταση να ε, αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί η ισότητα αυτό σημαίνει. Εφόσον έχω διαφορετικές καταστάσεις, πρέπει να έχω τη δυνατότητα, την ευελιξία και την πολιτική ικανότητα να λάβω υπόψη την ιδιαιτερότητά τους. Γιατί διαφορετικά αυτό το σύστημα το ε, φορολογικού ανταγωνισμό που εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί. Αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω μέσο για να διαβρωθούν οι αξίε. Γιατί διαφορετικά οι πιο αδύναμοι θα μείνουν πάντοτε πιο πίσω από του υπόλοιπου. Και συμφωνώ απόλυτα με του συναδέλφου από το ΙΝΕΣΕΝΤΗ και την ΚΟ ότι αυτή εδώ η γνωμοδότηση θα πρέπει να οδηγήσει σε τέτοιο, να, καταλήξει έτσι ώστε να στηρίξει αυτούς που δεν μπορούν να έχουν την πολυτέλεια του φορολογικού τουρισμού που άλλοι μπορούν να κάνουν επειδή έχουν τεράστιες πόρους για να πληρώνουν. Ε, και το λέω γιατί είμαι και εγώ ίδιος γιος ενός μικρού επιχειρηματίου και γι' αυτό το θέμα αυτό με διαφέρει πολύ και με παθιάζει. Ε, έχουμε λοιπόν μέχρι την 1η Οκτωβρίου για να ε, τελειοποιήσουμε το περιεχόμενο της ε, γνωμοδότησης και εγώ μέσω των συζητήσεων έχω, έχω οδηγηθεί μάλλον σε κάποιες τροπολογίες που θα καταθέσω και σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ξεκάθαρες οι απαντήσεις για όλες τις παρατηρήσεις σα. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών για αυτό το σχέδιο χρηματοδότησης είναι στην 1η Οκτωβρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι. Εντάξει, το καταλάβατε όλοι. Και τώρα θα έχουμε 4 λεπτά διάλειμμα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε ακριβώς στις 5. 4 λεπτά διάλειμμα. Sorry, I was slightly too long because I lost myself in the European Parliament. well, it could happen sometimes. Uh, if I may, welcome. Λοιπόν, καλώς ορίζω. Το ε, κύριο Πέτρο Σολμερίπ που είναι ε, θυμηματάρχης στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντικό το briefing, η ενημέρωση που θα μας κάνει για τις διαπραγματεύσεις του TTIP, όπως θα θυμάστε μάλλον. Βρισκόμαστε στο δέκατο γύρο επίσημων διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκε τελευταίος ήταν στις Βρυξέλλες 13 με 17 Ιουλίου του 2015 είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τον Ιούνιο του G7, οι ηγέτες, όχι της Γενικής Διεύθυνσης 7, του G7, μαζί με τους προέδρους ε, Τούσκ, Γιούνκερ και Ομπάμα, ε, έδωσαν σαφείς εντολές να ενταθούν οι συνομιλίες για το TTIP και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε όλους τους τομείς. Το ίδιο ε, ισχύει και για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών που ενέκρινε ε, τον Ιούνιο σχετική νομοθεσία για να δοθεί και επιπλέον πολιτική όθηση και να υποστηριχθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ήδη λοιπόν εκατέρωθεν του Ατλαντικού επιθυμούμε και εκφράστηκε αυτή η επιθυμία να προχωρήσουμε ταχύτερα. Και στις 8 Ιουλίου του 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διατλαντικό εμπόριο ε, και ε, τις επενδυτικές ε, σχέσεις, το TTIP. Για τους διαπραγματευτές λοιπόν και είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή η κατάσταση μετά το G7, μετά τις δικές μας συστάσεις και μετά το δέκατο γύρο διαπραγματεύσεων να μάθουμε πού βρισκόμαστε. Το λόγο έχει ο κύριος Σολμέρης για να μας ενημερώσει για το δέκατο γύρο διαπραγματεύσεων. Βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις <laughs> για τον ένατο ή για τον όγδοο γύρο βεβαίως μπορείτε να τις κάνετε. Δεν αφορά η συζήτηση μόνο τον τελευταίο γύρο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Γεια σας. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να σας ενημερώσουμε για τις διαπραγματεύσεις του TTIP. Η τελευταία ενημέρωση, αν δεν απατώμε, ήταν το Μάιο. Θα πρότεινα λοιπόν, αν συμφωνείτε Πρόεδρε, να σας δώσω μια γενική ενημέρωση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων που βρισκόμαστε και να κάνουμε και μερικά σύντομα ειδικά σχόλια για την ενέργεια και ε, για τις πρώτες ύλες, για τις διαπραγματεύσεις εκεί και ε, για το σκέλος των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων όπου συμμετέχω πολύ και εγώ στις διαπραγματεύσεις αυτές και είναι θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τις εργασίες της Επιτροπής σας. Γενική τώρα ενημέρωση όπως γνωρίζετε το TTIP είναι μια διαπραγμάτευση με πολλές προκλήσεις και από τότε που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δρά επικοδομητικά και ε, συνεργάζεται παντού. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις σε κατέρωθεν του Ατλαντικού από το Μάιο που είχαμε την τελευταία ενημέρωση και θα ήθελα να αφαιρθώ. όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ε, το νόμο για την προώθηση του εμπορίου και την αντίστοιχη αρχή που επιτρέπει στον πρόεδρο Ομπάμα να προχωρήσει με αυτό το θέμα. Προσπάθησε ε, ε, να ολοκληρώσει το ίδιο από πλευράς ειρηνικού το TPP, αλλά διαφώνησαν σε θέματα αυτοκινητοβιομηχανίας και γαλακτοκομικά με κάποιους από τους εταίρους τους του ειρηνικού. Ε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να επιληθούν τα αυτά ε, τα εκκρεμή ζητήματα. Για το TTIP ε, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία του Ειρηνικού. Θα πρέπει και το TTIP να προχωρήσει για να έχει πλήρη ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, ε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίθηκε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη πλειοψηφία και αυτό έδωσε και σημαντική πολιτική στήριξη στι διαπραγματεύσει. Τώρα έχουμε μια σαφή πολιτική πλατφόρμα για να πιέσουμε ε, για μια συνολική συμφωνία υψηλών προτύπων και προδιαγραφών. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ενέκρινε μια πρόταση για προστασία των επενδύσεων και ε, ένα σύστημα ε, δικαστηρίου λύσης των διενέξεων Βεβαίως με διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρότασης και των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερομένων. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΙΤΑ συνεδριάζει και στην ΙΤΑ κάποιοι συναδελφοί μου παρουσιάζουν την πρόταση αυτή εκεί. Θέλαμε αυτή την πρόταση να την φέρουμε και να την παρουσιάσουμε πρώτα και να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη πριν ε, την ολοκληρώσουμε και τη στείλουμε ως νέα πρόταση στις ΗΠΑ, Πολιτείες, στις διαπραγματεύσεις. Γενικός μας στόχος παραμένει να κλείσουμε με την παρούσα κυβέρνηση Ομπάμα και θέλουμε να κάνουμε παντού πρόοδους και έχουμε προτάσεις σε όλους τους τομείς και μέχρι τέλη του έτους μας ενδιαφέρει να έχουν κατατεθεί. Βεβαίως ε, θα πρέπει η ουσία να ε, είναι σημαντικότερη και όχι η ταχύτητα. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων θα αναθεωρηθεί από την Επίτροπο ε, Μάλστρομ και ε, αύριο μαζί με τον επικεφαλής ε, διαπραγματευτή των ΗΠΑ, Φρόμαν. Τα θέματα πρόσβαση στην αγορά επίσης ήταν καθόδη μέχρι τώρα και θα πρέπει να ανοίξουμε ένα δρόμο για να βρούμε πρόοδο και να επιτύχουμε για ε, τις υπηρεσίες, τις κρατικές προμήθειες και τις, τους δασμούς. Αυτά όλα συνδέονται και ε, χρειαζόμαστε μία σαφή συμφωνία για να διαπραγματευτούμε την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις γιατί υπάρχουν κάποιες ε, κρατικές ε, πολιτικές όπως το Buy America, να αγοράζει τα αμερικανικά προϊόντα και κάποιες διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση στους διαγωνισμούς στις δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ και θέματα που έχουν να κάνουν με την πρώτη ή τη δεύτερη προσφορά ε, σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτά πρέπει να λυθούν παράλληλα ε, κάθε στοιχείο που έχει να κάνει με την πρόσβαση στις αγορές. Επίσης έχουμε συνεργασία για το κανονιστικό πλαίσιο. Θέλουμε μια συμφωνία υψηλού επίπεδου ψηλών προδιαγραφών με απτά χειροπιαστά αποτελέσματα και να μην μειωθεί η σημερινή προστασία μας και τα επίπεδα που επικρατούν για το υπόλοιπο του έτους που απομένει ε, θέλουμε να προχωρήσουμε και να δούμε πώς μπορεί ο κάθε κλάδος να καταλήγει και κάθε συζήτηση. Στο πυλώνα των κανόνων θα πιέσουμε να ενταθούν οι προτεραιότητες, ε, οι δικές μας που είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις και η ε, ενέργεια και οι πρώτες ύλες ε, που είναι ένα θέμα στο οποίο θα επεκταθώ στη συνέχεια μετά τη γενική αυτή παρουσίαση. Επίσης υπάρχει και η δική μας πρόταση για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό θα κυριαρχήσει στον επόμενο γύρο, μη γύρους το διαπραγματεύσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, πλήρη υποστήριξη, η Επίτροπος, να συνεχίσει ε, τις διαπραγματεύσεις και τα κράτη-μέλη αν δείξουν και πολιτική υποστήριξη αυτό θα μας βοηθήσει κάνουμε προσπάθειες να κερδίσουμε και τη δημόσια συζήτηση ε, υπάρχει μια τεράστια πίεση για διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Γίνονται προσπάθειες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, για τη δημόσια συζήτηση, αλλά αυτό δεν είναι μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη. Θα πρέπει πολιτικοί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυβερνήσεις να βοηθήσουν. Ε, η Επίτροπος Μάνστομ είναι υπέρ της περισσότερης διαφάνειας και οι μόνες αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι προς μεγαλύτερη διαβάνεια, όχι μικρότερη. Έρχομαι τώρα στα θέματα ενέργειας και πρώτων υλών και στις σχετικές συζητήσεις, Πρόεδρε. Στο 10ο γύρο λοιπόν τον Ιούλιο είχαμε τεχνικές συζητήσεις που συνεχίστηκαν ε, παντού. Αυτές έγιναν με την επιφύλαξη υφισταμένων κεφαλαίων ε, για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει ακόμα πολιτική απόφαση από αυτόν. Στο μεταξύ θα πρέπει εμείς όμως να προοδεύσουμε, να δούμε ποια είναι τα συστατικά αυτά ε, μια ενδεχόμενη συμφωνίας εκεφαλαίου για την ενέργεια και τις πρώτες ύλε, για να διευκολύνουμε την πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί σύντομα είναι ευθυγραμμισμένη και με τα συμπεράσματα των G7 που μόλις εσείς Προέδρε αναφέρατε. Και τα συμπεράσματα αυτά του Ιουνίου ζητούν επιτάχυνση σε όλους τους τομείς και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε όλους τους τομείς και στην ενέργεια και στις πρωτεσίλες μέχρι τα τέλη του 2015. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης από την αρχή την ανάγκη να υπάρχει μια ισορροπημένη έκβαση και στο θέμα της ενέργειας και των πρώτων υλών και αυτό το κεφάλαιο δεν θα πρέπει μόνο να επικεντρώνεται στα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και θα πρέπει να λύσουμε τις δυσκολίες πρόσβασης ε, στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο των ΗΠΑ γιατί έχουν περιορισμούς στις εξαγωγές. Ένα τέτοιο κεφάλαιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για να υπάρχει ισόρροπη και βιώσιμη προσέγγιση. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του, το οποίο πάρα πολύ χρήσιμο τόνισε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τους ευρύτερους γεωστρατηγικούς λόγους που καθιστούν την ενέργεια και ε, τα, τα, τα, τις πρώτες ύλες απαραίτητα ως ξεχωριστό κεφάλαιο στο TTIP. Επανέρχομαι στο γύρο του Ιουλίου, συζητήσαμε θέματα πρώτων υλών έτσι, σε πολύ μεγάλη έκταση και διευρύνθηκε και το πεδίο ε, ε, όσων ενδεχομένως καλυφθούν στη συμφωνία και πώς θα πέσουν τα εμπόδια και οι φραγμοί που υπάρχουν στο εμπόριο πρώτων υλών, όχι τόσο πολύ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σε σχέση με τρίτες χώρες όπου μπορεί να έχουμε κοινά συμφέροντα. Επίσης, αναθεωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες συνεργασίας στην ενέργεια και στις πρωτοσύλλες και συμφωνήσαμε Συζητήσαμε μάλλον ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στη συμφωνία. Ο επόμενος γύρος θα είναι στο Μαγιάμι στις εβδομάδα της 19ης Οκτωβρίου για την ενέργεια και, τα ορυκτά, και τις πρώτες ύλες ε, μια εβδομάδα πριν στην Ουάσιγκτον, στις 12 Οκτωβρίου δηλαδή. Στόχος είναι να εστιάσουμε σε διάφορα θέματα που μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει και καθώς ε, προχωρούμε προς τα τέλη του έτους θα πρέπει να κινηθούμε προς την ολοκλήρωση των τεχνικών συζητήσεων για Ε, διάφορα στοιχεία που θα μπουν σε αυτό το κεφάλαιο για να διευκολυθούν και οι πολιτικές συζητήσεις ε, βάσει των συμπερασμάτων του G7. Από δύο λόγια ίσως ε, κλείνοντας για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως θα θυμάστε, το TTIP είναι η πρώτη συμφωνία FTA που διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες, όπου έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και συμφώνησαν και οι δύο πλευρές να υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ότι ένα τέτοιο κεφάλαιο θα πρέπει να εστιάζει σε τρία θέματα θέματα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ε, τη σύσταση μιας επιτροπής για τις μικρομεσαίες. Το πρώτο στοιχείο της συνεργασίας έχει προχωρήσει περισσότερο από τα άλλα μέχρι στιγμή στη διαπραγμάτευση. Ε, οικοδομούμε στην ε, υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Growth και των ομολόγων από πλευράς ΗΠΑ ειδική συνεργασία για θέματα που έχει να κάνει με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανταλλαγή πληροφοριών ακόμα υπολείπεται. Μένει δουλειά για να συμφωνήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος των πληροφοριών ε, που θα ανταλλάσσουμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μαθαίνουν περισσότερο για τις ευκαιρίες που θα τους δίνει αυτή η συμφωνία και να γνωρίζουν καλύτερα γενικότερα πώς λειτουργεί η αγορά τις Ηνωμένε Πολιτείε και δηλαδή πώς μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους εκεί. Από δική μας πλευράς έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται Export Help Desk ε, που βοηθάει για τις εξαγωγές και το χρησιμοποιούμε για τη δική μας αγορά, την εσωτερική. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει και ένα αντίστοιχο μέσο για τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις με την Αμερική. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα ε, στο μέτωπο εκεί των μικρομεσαίων και το τρίο ε, έχει να κάνει με ε, μια επιτροπή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προβλέπεται να συσταθεί. Ε, γιατί έχει σημασία αυτό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυσικά θα χρειαστούν να εποφελούνται από τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν από την συμφωνία. Δεν είναι μόνο ένα ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες, είναι γενικότερα συμφωνία. Οπότε θεωρούμε ότι ε, με μια τέτοια επιτροπή θα μπορούν να συνδέονται με τα άλλα στοιχεία της συμφωνίας και τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή υπάρχει το θεσμικό σκέλος της συμφωνίας και μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό πριν ολοκληρώσουμε γενικότερα την ε, συμφωνία στο σύνολό της. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία στοιχεία, τρει τομεί για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και στον 11ο γύρο θα εξακολουθήσουμε να ε, εργαζόμαστε από αυτόν τον Οκτώβριο. Και πρέπει να σα πω ότι σε σύγκριση με άλλου τομεί ε, έχει επιτελεστεί ήδη μεγάλη πρόοδο για τις ΗΠΑ, αλλά εκκρεμούν και άλλα ζητήματα που πρέπει να λυθούν και να ολοκληρωθούν. Προτείνω να σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, και βεβαίω με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Πολ Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να συζητήσουμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που να κερδίζουν όλοι, μια κατάσταση win-win. Και το θέμα Τη ενέργειας και των πρώτων υλών είναι κεντρικό για την Επιτροπή μας. Τι δυνατότητες υπάρχουν εξαγωγής ενέργειας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι γίνεται με τις άδειες και ο ενεργειακός χάρτης θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή και θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων αυτών. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με τη βιομηχανική πολιτική. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση της Volkswagen. 18 ε, δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμο έχει επιβληθεί. Είδαμε τα πρόστιμα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Google. Αυτά είναι ένα είδος φορολογίας αυτά τα πρόστιμα. Συζητήσαμε σήμερα το θέμα της εταιρικής φορολογίας. Εσείς πώς βλέπετε τα πρόστιμα αυτά. Και θα ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχει ε, το νομοθέτημα «Αγοράστε αμερικάνικα προϊόντα», «Buy American». Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ερώτησή μου είναι τι μπορούμε παραπάνω να συμπεριλάβουμε στην TTIP από ότι ε, στις ε, διακολύνσεις ε, που έχουμε στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και ζητώ συγγνώμη που μπούκαρα ενώ ήδη είχατε πάρει εσεί το λόγο. Καλωσορίζω την πρόοδο που είπατε ότι κάνετε στον τομέα των μικρομεσαίων. Μία από τις προκλήσεις στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένω γι' αυτό το θέμα ήταν η έλλειψη διαφάνειας στι ΕΠΑ όσον αφορά το νομοθεσία σε κρατικό επίπεδο και τους κανόνες που ισχύουν για το τομέα των υπηρεσιών. Τι είδους εργασία γίνεται ώστε να κατηγοριοποιηθούν και να καταγραφούν οι κανόνες και τα προδιαγραφές των ΙΠΑ. Τώρα, μιλήσατε για συνεργασία για τις πρώτες ύλες σε τέτοιες χώρες όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Ως Ήπειροι έχουμε τώρα νομοθεσία ή φτιάχνουμε νομοθεσία όσον αφορά τα όρυκτα των συγκρούσεων. Ε, είναι αυτό κομμάτι της συζήτησης όταν μιλάτε για πρώτες ύλες, γιατί είναι ένα τομέα που θα μπορούσαμε να βρούμε ένα είδος ε, στάνταρ χρυσού ε, να αναπτύσσεται, αν υιοθετούσαμε δηλαδή κοινού κανόνες σε αυτό το τομέα. Έπειτα γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μόλις υιοθέτησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ερευνητικό ε, για πολιτική και για θετική έρευνα όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια. Ελπίζουν ότι η ΕΠΑ θα μπορέσει να ηγηθεί του κόσμου σε αυτές τις ε, ενέργειες, ενώ η Ευρώπη είχε ανέκαθεν την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα. Εσεί αναφέρατε ερευνητικά προγράμματα. Τι είδους συνεργασίες ε, κάνετε ώστε να μην χάσουμε το στάτους μας στην αγορά όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και επάρκεια και τη σχετική τεχνολογία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα όσα ακούσαμε και μάλιστα δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω όταν δηλώσατε ότι χρειάζεται πολιτική στήριξη από τα κράτη-μέλη ώστε να κερδίσουμε τους συμπολίτες μας. Εγώ προέρχομαι από την Αυστρία και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολο το πράγμα και ήμουν ανέκαθεν υπέρ μιας προσπάθεια επικοινωνιακής που θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Ως προς αυτό το θέμα παρακολουθούμε τις νέες προτάσεις σε σχέση με της, ε, ε, το Δικαστήριο Επενδύσεων και επίσης ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται υπόψη μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αυτή τη νέα πρόταση και ότι θα έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας επόμενο ομιλητή, εξ της η κυρία Λόπε. Βερβέγουα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ενημέρωση για αυτή τη δέκατο γύρο διαπραγματεύσεων. Εγώ στην πράξη θα ήθελα να σας διαβιβάσω κυρίως ανησυχίες που έχουμε από πλευράς της ομάδας μας, της ΓΟΕ. Στην πράξη, οι ανησυχίε που έχουμε είναι ότι ανοίγει η πόρτα ώστε οι ΙΠΑ να επιβάλλουν την απελευθέρωση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ε, μία παράλυση προβλέπεται για τις εργαστικές νομοθεσίες αλλά και τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες ε, έτσι ώστε να μην ε, ε, ενισχυθεί ε, ο ανταγωνισμός με μια χώρα που δεν υπάρχουν αυτές οι διατάξεις όπως είπα. Ανησυχώ πολύ με για τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Το ΡΕΦΙΤ θεωρώ ότι προβλέπει τα όσα προβλέπει τι τύπος όσον αφορά την απελευθέρωση και την απορρίθμιση. Το ίδιο για τις βιομηχανίες και για τους ε, τομείς χαμηλής ε, προστιθέμενες αξίες όπως ε, οι βιομηχανίες που έχουμε στην Ισπανία και όπου είπα, έχουν ε, ανταγωνιστικότητα μέσω της υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Φοβούμεθα ότι θα εξαφανιστούν βιομηχανίες όπως η χημική ή η αυτοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης το πρόβλημα των βιομηχανιών όπως η αγροδιατροφική ή η αγροβιομηχανική όπου ε, οι υποχωρήσεις θα, οδηγούσε, θα οδηγούσαν στο μεγαλύτερη ακόμα εξάρτηση από τις εισαγωγές, από τις είπα, εις βάρος της τοπικής μεταποίησης ή στην εξαφάνιση της ίδιας μας της βιομηχανίας από τη στιγμή που θα εξαφανιστούν οι δεσμοί της με την ε, επικράτεια, με τις συγκεκριμένες περιφέρειες. Υπάρχει επίσης ε, ο κίνδυνος του μονοπωλιακού ελέγχου της γνώσης, γιατί έτσι Ανησυχούμε ότι θα διδικοποιηθεί η τεχνολογική βελτίωση στα χέρια κάποιων λίγων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ραιλή η Ο κύριο Μπορέλη, εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Δηλαδή, στι τεχνικέ διαπραγματεύσει μπορεί να υπάρξουν ε, παρεμβάσει με το θέμα τη Κίνα, δηλαδή την ενδεχόμενη αναγνώριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση του καθεστώτο οικονομία αγορά και τη συμφωνία του TTIP. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ο Κρίστιαν. Κρίσιαν, είσαι ο επόμενος στον κατάλογο. Είναι η ευκαιρία σου. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν μόνο οι συντονιστέ. Έχω μια απλή ερώτηση όσον αφορά τα αριθμιστικά ζητήματα και την ε, τυποποίηση. Διαβάζουμε πολύ προσεκτικά τη ε, έγγραφα της διαπραγμάτευσης που δείχνουν σχετικά υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά έλλειψη λες λεπτομέρειες μπορεί να είναι ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα. Πόσο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσει σε αυτό το τομέα. Από ό,τι καταλάβαμε δεν υπάρχει ακόμα εντολή από πλευρά των ε, ε, μετόχων όσον αφορά την ρύθμιση τυποποίηση των, του αντίστοιχου οργανισμού τυποποίησης μάλλον στις, ε, στις ΕΠΑ, ενώ έχουμε ε, την περασμένη εβδομάδα ακούσει τους επόπτες, ε, τις εποπτικές αρχές και έλεγαν ότι δεν υπάρχει μεγάλη συντονισμό ανάμεσα στο κεντρική εποπτική αρχή και τα ρυθμιστικά, εθνικά όργανα για αυτό το θέμα γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα. Πού βρίσκεται λοιπόν, πού είναι η εξέλιξη, πού βρίσκεστε σε σχέση με το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπυράκη, επόμενη μιλήτρια. Thank you, Chair. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση που μας κάνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εκ μέρους της Επιτροπής, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να γεφυρώσει την έλλειψη ε, ενημέρωσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά το IFTS, ε, τι είδους φορέα θα έχουμε, θα είναι ένας φορέας ad hoc και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Σμαρτάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ενημερώνει για την κατάσταση των προγραμμάτων. Εδώ είμαι εδώ. Στις Ηνωμένε Πολιτείες Όλο και περισσότερο Αμερικανοί αντιτίθενται σε αυτή τη συνθήκη ε, και πολιτικοί και πολίτες απλοί. Το ίδιο ισχύει και για τούτη την όχθη του Ατλαντικού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αισθάνονται ότι θα βγουν χαμένοι. Οπότε έχω και εγώ μια πολύ απλή, ίσως απλοϊκή ερώτηση. Πιστεύετε ακόμα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ε, μήπως να σταματήσουμε εδώ πέρα να περιορίσουμε και τις ζημιές, όπως ορισμένοι προτείνουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την τεχνική ενημέρωση που μας έκανε και που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να αποδεσμεύσουμε την τεχνική ενημέρωση από την εξέλιξη του πολιτικού πλαίσιου. Πριν από λίγο ο ο συνάδελφος Μαρτέ το ανέφερε και εκείνο. Και τι πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλα δυνητικά πλεονεκτήματα και την Ευρώπη και τον κόσμο που θα απορρέψουν από μια τέτοια συμφωνία. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να το αξιοποιήσουμε. Για παράδειγμα, διάσκεψη κορυφής ενέργεια-κλίμα. Και το τι θα προκύψει από αυτή τη διάσκεψη κορυφής θα είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική συμφωνία ανάμεσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν προετοιμαστούμε όμως όπως δει, μπορεί όντως ε, οι ΙΠΑ να προηγηθούν ε, και, στο θέμα της ενέργειας, ε, της και στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε άλλη φάση κρίση στη Λατινική Αμερική και στο οικονομικό πρότυπο, μοντέλο της Λατινικής Αμερικής. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την TTIP ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα φάση στο Μερκοσούρ πριν λίγο καιρό αυτές οι κυβερνήσεις έδωσαν την όθηση στην ε, εξέλιξη αυτών για αυτές τις χώρες. Πολλές φορές η όθηση δίνεται με βάση ε, το κατά πόσο οι περιστάσεις βοηθούν και θα πρέπει τώρα οι δικές μας κυβερνήσεις να δώσουν αυτή την όθηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Η ερώτησή μου είναι μάλλον πολύ απλή ποιο θα είναι το τέλος των διαπραγματεύσεων, πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε και ποιο θα είναι το γενικό χρονοδιάγραμμα μετά την, ε, το λεγόμενο τέλος των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα δηλαδή να ξέρω πότε θα ξεκινήσει να ισχύει ε, η όλη συμφωνία. Δεύτερη ερώτηση. Νομίζω ότι το ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια συνεχίζει να μας ενδιαφέρει και βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας. Και τρίτο θέμα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, άνοιγμα των συνόρων για το εμπόριο. Εξαγωγές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έχουν τα πράγματα και Σημείο 4. Πληροφόρηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κάποιος αναφέρθηκε στις δημόσιες συμβάσεις. Κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μάλλον είναι και το πιο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι καταλάβαμε, Αναφέρθηκαν κυρίως τεχνικά ζητήματα, παρόλα αυτά μερικά είναι σημαντικά και σχετίζονται με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Έχετε το λόγο να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω από την ερώτηση του κύριου Μαρτά. Γιατί είναι θεμελιώδης ερώτηση για τη συζήτησή μας. Ναι, σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο καλά μπορώ. Ε, να γνωρίζετε όμως ότι είμαι ο κύριος διαπραγματευτής για το θέμα της ενέργειας και όχι για το σύνολο της συμφωνίας. Η απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Μαρτά είναι σαφής από τη δική μας την πλευρά. Ναι, πιστεύουμε ότι πρόκειται για θεμελιώδους σημασίας συμφωνία. Πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε με τη σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας TTIP και πιστεύουμε ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται μια τέτοια συμφωνία σήμερα περισσότερο από ποτέ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο, ο Επίτροπος και όλες οι υπηρεσίες εργάζονται σκληρά νυχθημερών για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να περάσω στην δική σας ερώτηση, διότι πιστεύω ότι είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας. Ποιο θα είναι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Σας είπα ότι για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις Μάλλον όταν μιλάμε για το τέλος των διαπραγματεύσεων θα μιλάμε για την ολοκλήρωση του έργου των διαπραγματευτών, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και από τις δύο πλευρές από τα αρμόδια όργανα και να εγκριθεί. Στη δική μας περίπτωση, όπως γνωρίζετε, τα αρμόδια όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν, όπως γνωρίζετε. Που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, με την εξέταση, με την μετάφραση του κειμένου προτού να προχωρήσουν τα θεσμικά όργανα στην επί της ουσίας εξέταση. Στόχος μας είναι λοιπόν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Ομπάμα. Αυτός ο χρόνος όμως διαφέρει από τον χρόνο που θα πετηθεί για την θέση σε ισχύ της συμφωνίας και η ΠΙΑ μας έχει δείξει ότι απαιτείται αρκετό χρόνος λόγω ε, των διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμοστούν προτού να μπορεί να τεθεί σε ισχύ ε, μια συμφωνία. Μάλλον ε, ένας χρόνος ή δύο χρόνια θα χρειαστούν. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στη σημασία να υπάρχει ε, ειδικό κεφάλαιο για την ε, ενέργεια και προσπαθούμε να σημειώσουμε όσο γίνεται περισσότερη πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο για να συζητήσουμε ε, το ERM την ενέργεια δηλαδή και τις πρώτες ύλε. Και συζητούμε με τις ΗΠΑ τη συμπερίληψη ενός τέτοιου κεφαλαίου. Και εφόσον συζητήσαμε στο πλαίσιο των G7 να εντατικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να έχουμε κοινή κατανόηση για κάθε κεφάλαιο πριν το τέλος της χρονιάς, πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι και το χρονοδιάγραμμά μας ε, για την πρόοδο που θα πρέπει να σημειωθεί στον ε, τομέα της ενέργειας ε, και των πρώτων υλών. Όσον αφορά τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, ο κύριος Ρούπιχ έθεσε κάποιες ερωτήσεις. Ρωτήσατε αν θα εφαρμοστεί ο ενεργειακός χάρτης στο πλαίσιο του κεφαλαίου ε, για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες ε, στη Συμφωνία TTIP. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε συνυπογράψει τον ενεργειακό χάρτη, ε, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι. Οι προτάσεις μας στη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται σε αρχές που έχουν αναπτυχθεί στην συνθήκη του ενεργειακού χάρτη συζητάμε με τις, Ηνωμένε Πολιτείε ώστε να έχουμε διατάξεις που να βασίζονται στις αρχές αυτές. Ένα παράδειγμα είναι ο χώρος διέλευσης, διαμετακόμισης. Επίσης, τονίσατε τη σημασία του νομοσχεδίου «Αγοράστε Αμερικανικά προϊόντα» «Buy American». Αυτό μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο των ε, δημοσίων συμβάσεων. Αναφέρθηκα στην ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους τομείς όσον αφορά την ε, πρόσβαση στην αγορά, όσον αφορά δηλαδή τις υπηρεσίες ε, και τα προϊόντα στον τομέα των δημοσίων προμηθειών στον τομέα αυτών. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα του νομοθετήματος αυτού και θα πρέπει να τα συζητήσουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Επίσης, μας ρωτήσατε τι παραπάνω θα μπορούσαμε να έχουμε στη συμφωνία αυτή, πέρα δηλαδή από όσα έχουμε στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Και η ενέργεια και οι πρώτε ύλε από τη μία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την άλλη αποτελούν παραδείγματα του τι μπορεί να προσθεθεί στους γενικούς κανόνες που ισχύουν. Παρότι οι κανόνες του που ισχύουν για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες δεν καλύπτουν ε, όλα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στον τομέα αυτών. Αυτή λοιπόν θα ήταν μια χρήσιμη προσθήκη, όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν αναφέρονται στους πολυμερούς κανόνες. Στους πολυμερείς κανόνες. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που σχεδιάζουμε διατάξεις που σχετίζονται ειδικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, κύριε Κίρτον Τάρλινγκ, σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας ε, των επενδύσεων. Σχετίζεται και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και την δημιουργία εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε για την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας. Ελπίζουμε δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε και σε επίπεδο μεμονωμένων πολιτιών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτόν. Αναφερθήκατε και στα, στην νομοθεσία για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Οι Ηνωμένε Πολιτείες υιοθέτησαν κάποιες διατάξεις που απαιτούν δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ορυκτά από τις περιοχές των μεγάλων λιμνών, από την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και θα ξεκινήσει τριμερή διάλογος ε, με την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου. Αυτό δεν συζητιέται άμεσα στις διαπραγματεύσεις TTIP και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι και εμείς και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε σχετική νομοθεσία που βασίζεται στις κατευθυντές γραμμές του ΩΣΑ. Έχουμε λοιπόν κοινή βάση το θέμα αυτό. Δεν είναι παρόμοιες σε όλα τα σημεία οι νομοθεσίες μας. Ούτε θα ήθελα να αναφερθώ στο ποιο θα μπορούσε να είναι το πιθανό αποτέλεσμα της νομοθετικής εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών, αλλά οι νομοθεσίες μας έχουν τον ίδιο στόχο και θα βασίζονται στο ίδιο διεθνές πλαίσιο του ΩΣΑ. όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. είναι κάτι που θα μας αποσχολήσει στο πλαίσιο της ενέργειας και των πρώτων υλών για να πετύχουμε ισορροπημένο αποτέλεσμα. Είναι ένας τομέας όπου είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι, όπως είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Αναφέρομαι στην ε, ανάπτυξη προτύπων ενεργειακής απόδοσης και δοκιμών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, αν ε, θέλουμε να κάνουμε κάτι κοινό στον τομέα αυτόν. Νομίζω ότι εκφράστηκαν ανησυχίε από την κυρία Λόπες Περμέχο. για το επίπεδο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα προσπαθούμε να είμαστε σαφείς στο θέμα αυτό και θα το επαναλάβω και σήμερα. Τίποτα στη συμφωνία αυτή δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο προστασίας που ε, έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά αναφέρεται το παράδειγμα των χημικών, όπου έχουμε τον κανονισμό REACH στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή Είπαμε ότι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γνωρίζοντας ότι έχουμε διαφορετικό σημείο κίνηση. Εμείς έχουμε τη δική μας νομοθεσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τη δική τους. Έχουν διαφορές οι νομοθεσίες αυτές και στόχος δεν είναι να αλλάξουμε τίποτα στην νομοθεσία REACH. Και αυτό ισχύει για όλους τους τομείς. Νομίζω επίσης ότι τέθηκε μια ερώτηση που δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις αυτές καθ' αυτές για την Κίνα και για το ε, καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Δεν υπάρχει εδώ άμεση σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Όσον αφορά την αξίωση της ε, Κίνας να αποκτήσει καθεστώς ε, οικονομίας της αγοράς. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις περί τυποποίησης, ε, νομίζω ότι ο κύριος Σίλερ έθεσε ερώτηση για το θέμα αυτό. Εργαζόμαστε εδώ σε διάφορα επίπεδα. Ε, έχουμε το τεχνικό επίπεδο, έχουμε τα φυτιο θέματα, όπου έχουμε δύο τελείως διαφορετικά συστήματα και μετά έχουμε τομεακά θεματολόγια για διάφορους τομείς. Όπως είναι η συνεργασία πάνω σε μελλοντικού κανονισμούς, για παράδειγμα. Εδώ το αποτέλεσμα ποικίλει ανάλογα με τον τομέα. Σε κάποιους τομείς έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Τα υφάσματα είναι άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς δηλαδή όπου έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπου θα πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος. Επίσης θέθηκε μια ερώτηση από την κυρία Σπυράκη σχετικά με το δικαστήριο επενδύσεων που προτάθηκε. Προσωπικά δεν είμαι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Με ρωτήσατε εάν είναι ad hoc δικαστήριο. με τη διαπραγματεύση TTIP ε, σκοπός είναι να δημιουργηθεί δικαστήριο επενδύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από τους δικαστές το 1 τρίτο θα είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1 τρίτο πολίτες ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και το τελευταίο τρίτο πολίτες τρίτων χωρών. Και θα μπορούσε το δικαστήριο αυτό να εξετάζει τις ε, περιπτώσεις ε, προστασίας επενδυτών που θα υποβάλλονται. Αυτό λοιπόν το δικαστήριο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων TTIP. Θα συζητήσουμε και με άλλους εταίρους μας, ώστε πιο μακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί ένα διεθνές δικαστήριο στον τομέα αυτών. Ξεκινώντας όμως από τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Uh, I've tried to... Προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν ξέχασα κάτι, ευχαρίστως θα συζητήσω μαζί σας διμερώς. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, ποιος δεν είναι ικανοποιημένος με την απάντηση που έλαβε. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος, ε, διότι δεν ε, απαντήθηκε το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Κύριε Μαρτά, ήταν σαφής η απάντηση στην ερώτησή σας και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης ε, πιστεύει στις διαπραγματεύσεις και στην τελική σου επιτυχία. Ε, έχετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας επαναλαμβάνει την επίσημη ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι άλλο να πει, αλλά προσωπικά εσείς ως διαπραγματευτής το πιστεύετε ότι θα το φέρετε εις πέρας αυτό. Φυσικά και το πιστεύω, λοιπόν και μπορεί να είστε βέβαιος ότι το πιστεύω κράδαντα. Πρόεδρε, συγγνώμη, εσείς είπατε ότι μείνατε δυσαρεστημένος για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Θα ήθελα να σαφής, ίσως δεν ήμουν μέχρι στιγμής. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την ενέργεια και τις πρώτες ύλε, συζητούμε διάφορα θέματα. Και υπάρχουν δύο ζητήματα που συζητούμε με δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις διμερείς μας ε, σχέσεις επενδυτικές και τις εμπορικές Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε και το δεύτερο σκέλος είναι κάποια ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με διμερείς δυσκολίες αλλά με κάποια θέματα που θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις του TTIP θα μπορούσαν να καταλήξουν σε γενικότερους παγκόσμιους κανόνες ενδεχομένως όπως είπε και ο κύριος Ρουμπίχ στον ΠΟΕ υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση για να αναπτύξουμε κάποιους κανόνες για θέματα τα λεγόμενα του 21ου αιώνα. Λοιπόν, για το πρώτο σκέλος αυτής της εξίσωσης ε, που είναι οι διμερείς σχέσεις και τα προβλήματα και τριβές που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση στις πρώτες ύλες ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, κυρίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και αυτά τα ε, έχουμε βάλει στο κέντρο των διαπραγματεύσεων. Και να είστε βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας όλα αυτά. Βεβαίως, τώρα ικανοποιήθηκα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σορμελή για τις εξηγήσεις σας και με χαρά να σας ξαναδούμε, να μας πείτε για τον επόμενο γύρο και να μας ξανάρθετε. Λοιπόν, λήξεις, ραντεβού αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.